Okay. Uh, good day everybody. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα γυρίσω στα σουηδικά. Παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας για να ακούσετε τη μετάφραση. Uh, λοιπόν, θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους στην τελευταία συνεδρίαση του έτους. Πρώτο σημείο της ημερησίας διατάξεως, έγκριση της ημερησίας διάταξης. Έχει διανεμηθεί νωρίτερα, αλλά υπάρχουν κάποιες αλλαγές και πιο συγκεκριμένα το σημείο 15 θα το συζητήσουμε μετά το σημείο 4. Και επίσης και το 7 θα έρθει μετά το σημείο 4 και μετά το 15. Ενώ το σημείο 5 θα το συζητήσουμε αύριο μετά το σημείο 14. Ενώ το σημείο 18 θα συζητηθεί αύριο μετά το σημείο 5. Εγκρίνεται. Ωραία, ευχαριστώ. Περνούμε στο σημείο 2, ανακοινώσεις του Πρόεδρου. ανακοινώσει του Πρόεδρου. Α, μας προσφέρουν καφέ. Μισό λεπτό λοιπόν. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι θα υπάρξει ένα εργαστήρι για το MFF την 5η στις 27 Ιανουαρίου το πρωί. Και αυτό θα αποτελέσει μέρος της συνεδρίασης της Επιτροπής αυτής. Το πρόγραμμα βεβαίω θα σας διανεμηθεί. Θα ήθελα επίσης με την ευκαιρία αυτή να πω ότι η Καρολίνα Φόκ ε, δυστυχώς μας αφήνει, ε, δούλευε στη γραμματεία, μας ε, φεύγει λοιπόν τέλος Ιανουαρίου. Νομίζω ότι θα στεναχωρηθούμε πολύ εξημών με την αναχώρησή της, διότι η συμβολή της ήταν πολύτιμη. Ε, μας άρεσε ο τρόπος που εργαζόταν, ο αναλυτικός τρόπος, ο μεθοδικός. Λυπούμαστε λοιπόν που δεν θα είναι μαζί μας πλέον. Εγώ ε, στεραχωριέμαι ιδιαίτερως διότι δουλεύω μαζί της επί σειρά ετών. Ξέρω ότι είναι πολύ ταλαντούχα με πολλά προσόντα, αλλά ταυτόχρονα είμαι και ευτυχής για αυτήν και την οικογένειά της διότι είναι δική τους επιθυμία αυτή η μεταβολή πηγαίνει στη Σουηδία βρήκε μια δουλειά στη Σουηδία και θα δουλέψει εκεί Κάθε επιτυχία λοιπόν στη νέα σου καριέρα και ευχαριστούμε πολύ για όσα έκανες για την επιτροπή αυτή Eh, Παίρνουμε τώρα στο σημείο 3. Ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Έχει διανεμηθεί το κείμενο και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εικάζω ότι μπορούμε να ε, τα δεχθούμε. Και περνούμε στο σημείο 4 ανταλλαγή απόψεων με τον Επίτροπο Άντορ, Επίτροπο αρμόδιο για την απασχόληση, της κοινωνικής υποθέσεις και την ένταξη. Ο κύριος Άντορ έχει ένα πολύ περιορισμένο πρόγραμμα και πρέπει στις 4 να βρίσκεται σε μια άλλη συνεδρίαση. Συνεπώς η ανταλλαγή απόψεων θα πρέπει να είναι πολύ σύντομη. Θα πρότεινα οι συντονιστές Ε, να να έχουν το λόγο για δύο λεπτά και όλοι οι υπόλοιποι για ένα λεπτό ή τριάντα δευτερόλεπτα ή τα υπόλοιπα μέλη ένα λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει και ο κύριος Σάντορ το χρόνο να απαντήσει. Ο κύριος Κονίλσεν. Κοιτάξτε, είναι πολύ αυστηροί αυτοί οι κανόνες, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, θα δώσω το λόγο στον κύριο Άντορ. Σα ευχαριστούμε που είχατε την ευγενή καλοσύνη να έρθετε. Είχατε καιρό να έρθετε σε εμά. Λοιπόν, έχετε το λόγο αμέσω. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, χαίρομαι που είμαι μαζί σα σήμερα Γνωρίζω μερικούς και μερικές από εσά, ιδιαίτερα όσους ε, δραστηριοποιούνται σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό που βρισκόμαστε βέβαια και σε αυτή την ομιγύρη, γιατί η ισότητα των δύο φύλων στην πολιτική απασχόληση και την κοινωνική πολιτική ε, είναι προαπαιτούμενο για να εξασφαλίσουμε κοινωνική ισότητα αλλά και ε, οικονομική ευημερία. Υποστηρίζω λοιπόν τι προσπάθειές σα να εξασφαλίσετε ότι με γυναίκε και άντρε επωφελούνται εξίσου από τι οικονομικέ ε, ευκαιρίε και ότι προσπαθείτε ε, να μειωθούν και να εξαφανιστούν τα, μεταξύ, τα, οι διαφορές μεταξύ άνδρων και γυναικών. Έχετε συνεισφέρει πάρα πολύ στην ε, πολιτική ατζέντα ε, της ε, τρέχουσας οικονομικής κρίσης που όπως γνωρίζετε πολύ καλά ακόμα δεν έχει τελειώσει. Τελευταία, αναλύουμε τις κοινωνικές επιπτώσεις αυτής της κρίσης ιδιαίτερα εστιαζόμενοι στο ποιοι είναι οι ανεργοί ε, σε ό,τι αφορά το αν είναι γυναίκες ή άντρες ε, και την ηλικία τους. Όμως υπάρχουν και άλλες ε, πτυχές που είναι εξίσου σημαντικές με τις, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές τους επιπτώσεις. Για παράδειγμα, ποιες, τι τύπους δουλειές χάθηκαν, ε, σε τι κατάσταση βρισκόνται τα νοικοκυριά στα οποία συμμετέχουν αυτοί οι άνθρωποι κλπ. Οι κοινωνικέ επιπτώσει των εξελίξεων στην αγορά εργασία διαφέρουν ε, πολύ συχνά ανάλογα με το αν οι δουλειέ που χάθηκαν ήταν πλήρω μερική απασχόληση, αν ήταν ε, υψηλόμισθε ή χαμηλόμισθε, αν οι άνεργοι ζούσαν μόνοι του ή σε οικογένεια, αν ήταν οι μόνοι που είχαν εισόδημα στο νοικοκυριό ή όχι κλπ. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι κυρίως οι γυναίκες ανήκουν στις πιο ευάλωτες κατηγορίες. Υπ' αυτή την έννοια, πολύ πρόσφατα διάβασα την έκθεση του 2012 του, της Παγκόσμιας Ανάπτυξης για την ισότητα των διαφύλων και την ανάπτυξη που λέει ότι το πλεονέκτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά την ισότητα μεταξύ των Διοφύλων έχει διαβρωθεί. Οπότε αυτή η περιοχή πλέον μοιάζει πολύ περισσότερο στον υπόλοιπο κόσμο. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ενδεχομένε συνέπειε αυτή ε, τη δήλωση στην ε, διαμόρφωση πολιτική. Αν η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων δεν ενσωματώνεται στι πολιτικέ, θα πρέπει να πληρώσουμε πολύ ψηλό τίμημα εξαιτία των ε, δραματικών δημογραφικών αλλαγών και από την αυξανόμενη ανάγκη σε ό,τι αφορά θέσει εργασία. Γι' αυτό το λόγο πρέπει τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν υπόψη την ισότητα των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα και πολύ σοβαρά. Τώρα, πρωτοβουλίε τη ε, Κομισιόν σε ό,τι αφορά το, την διάσταση του φύλου. Ε, ε, σε, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Παρόλο ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένο στόχος για την απασχόληση των γυναικών στην στρατηγική του 2020, ε, αναφέρεται ρητά ότι το, ο στόχος είναι 75% απασχόληση στην η ε, ομάδα 20 64 ετών μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής των γυναικών. Αυτή τη στιγμή οι γυναίκες, τις γυναίκες δεν τις, δεν τις χρησιμοποιούμε επαρκώς. Ε, είναι ένα δυναμικό το οποίο δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί. 4 στους 5 που βρίσκονται στην αγορά εργασίας, 4 στους 5 άντρες είναι στην αγορά εργασίας, ε, ενώ το 1 τρίτο των γυναικών δεν είναι καν στον ενεργό πληθυσμό. Θέματα ε, είναι στο κέντρο του, ήταν στο κέντρο του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου και στην έκθεση ετήσιας ανάπτυξης 2011 και στο, στα συμπεράσματα του, του Συμβουλίου Απασχόλησης του Μαρτίου αναφέρονται σε μέτρα για να ενισχύσουμε την ε, απασχόληση των γυναικών. Λένε ότι τα φορολογικά στήματα και συστήματα κινήτρων θα πρέπει ε, να ε, βοηθούν το, το δεύτερο εισόδημα του κάθε νοικοκυριού που είναι κυρίω γυναίκε. Επίση, γονικέ άδειε, ευέλικτε μορφέ εργασία και μονάδε φροντίδα παιδιών ε, θα πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία. Το συμπέρασμα που βγαίνει από το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να υλοποιήσουν μια ε, συνολική πολιτική, ένα συνολικό μείγμα πολιτικών για να αντιμετωπίσουν τι διαφορέ μεταξύ φύλου σε ό,τι αφορά την απασχόληση. Ε, οι καταχώρα ε, ε, μάλιστα, το έλαβαν αυτό υπόψη τον Ιούνιο 2011, ήταν για συγκεκριμένα οκτω κράτη-μέλη. Οι συστάσει προβλέπουν ε, προσβάσιμες και οικονομικές ε, υπηρεσίες ε, φροντίδας παιδιών, μείωση των αντικινήτρων, φορολογικών αντικινήτρων, πιο ευέλικτες μορφές εργασίας και αντιμετώπιση του, της διαφοράς αμοιβή. Στο σύμφωνο Europlus, τρία κράτη-μέλη μάλιστα, ανέλαβαν, ε, ανέλαβαν περισσότερες ε, πιο προχωρημένες δεσμεύσεις ό,τι αφορά την, τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών. Σίγουρα ε, και πολλά άλλα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν παρόμοιες προσπάθειες. Η έκθεση φορολόγηση του 2012, του, του πακέτου για την ετήσια έκθεση ανάπτυξη του 2012, επαναλαμβάνει την ανάγκη να ξαναδιαμορφώσουμε τα φορολογικά συστήματα έτσι ώστε να διευκολύνουμε την συμμετοχή του δεύτερου εισοδήματο του καθηγητικού κυρίου και να ε, καταργήσουμε τις, ε, τα φορολογικά αντικίνητρα που υπάρχουν. Ε, Ω συμπέρασμα, το θέμα του φίλου ε, ήταν πολύ παρόν στο πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο και θα εξακολουθεί να είναι ψηλά στην πολιτική ατζέντα στο δεύτερο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η Κομισιόν παρακολουθεί προσεκτικά τις ε, δράσεις που αναλαμβάνουν τα κράτη-μέλη ε, για την υλοποίηση των συστάσεων σε αυτόν τον τομέα. Μια αξιολόγηση της ε, κατάστασης της εφαρμογής αυτών των συστάσεων θα μας δώσει τη βάση για τις καταχώρα συστάσεις του 2012. Τώρα, τα οικονομικά ε, χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να υποστηρίξουν τα προγράμματα ισότητας ε, των δύο φύλων γιατί βρίσκονται στο πυρήνα του κοινωνικού, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και θα παραμείνουν και μετά το 2013. Ε, μια ε, συνολική σφαιρική αξιολόγηση που ολοκληρώθηκε στην αρχή του 2011 απέδειξε ότι ε, υπάρχει ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία στην υποστήριξη του κοινωνικού ταμείου προ προς την πολιτική ισότητα δύο φύλων. Η συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου ήταν πολύ σημαντική, για παράδειγμα στην υποστήριξη για τη δημιουργία ενός, ε, μιας ε, αυτόνομης πολιτικής για την ισότητα των και την ανάπτυξη δεξιότητων των γυναικών και στην εφαρμογή δράσεων ε, όταν δεν υπάρχουν επαρκή κονδύλια στον εθνικό προπολογισμό. Όμως αυτή η αξιολόγηση επίσης κατέδειξε και μερικές δυσκολίες και περιορισμούς στο, στον τρέχοντα προγραμματισμό. Για παράδειγμα, ε, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση ε, των δράσεων που εστιάζονται στο φύλλο ε, και περισσότερη εφαρμογή μαλακών μέτρων, ήπιων μέτρων. Η αξιολόγηση απέδειξε ότι επίσης δεν υπάρχει σαφής κατανόηση τι σημαίνει mainstreaming σε ό,τι αφορά το φύλλο. Ε, στο ρυθμιστικό πακέτο που υιοθετήθηκε σε 6 Οκτωβρίου η Κομισιόν συμπεριέλαβε μια σειρά από διατάξει που θα ενισχύσουν τη συνεισφορά των διορθωτικών ταμείων και συγκεκριμένα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την βελτίωση τη ισότητα των δύο φύλων. Ε, το προσχέδιο του Γενικού Κανονισμού καθορίζει σαφώ την αρχή του mainstreaming ε, του, με βάση το φύλλο για όλα τα διορθωτικά ταμεία. Απαιτεί επίση ε, η σύμβαση εταιρική σχέση και τα, και επιχειρησιακά προγράμματα να περιλαμβάνουν συγκεκριμένε λεπτομέρειε για τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή αυτή τη αρχή. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό του Κοινωνικού Ταμείου, οι προτάσει τη Κομισιόν καθιστούν σαφέ ότι τα κράτη-μέλη θα προγραμματίσουν και θα εφαρμόσουν συγκεκριμένε δράσει. Συγκεκριμένε δράσει με στόχο να προωθηθεί η ισότητα μεταξύ άνδρων και γυναικών. Με άλλα λόγια, κάθε κράτο μέλο θα προωθήσει την ισότητα των δύο φύλων με την ε, βοήθεια του Κοινωνικού Ταμείου μέσω μια διτή προσέγγισης του mainstreaming και συγκεκριμένων δράσεων. Επιπλέον, το 2012 το πρόγραμμα προόδου θα συνεχίσει τις, ε, ήδη, τις δραστηριότητες και θα ε, προσθέσει και κάποιες καινούριες. Για παράδειγμα, πρώτον, ε, ο τομέας της, ε, του προγραμματισμού, του σχεδιασμού ε, πολιτικής και νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση συγκεκριμένα στοιχεία. Εκεί χρειαζόμαστε συγκεκριμένα στοιχεία που θα μας επιτρέψουν να έχουμε στα χέρια μας στατιστικές και δείκτες. Δεύτερον, αποτελεσματική πληροφόρηση και διαμερασμό της γνώσης. Νέες δραστηριότητες που αφορούν ε, ισότητα των εισοδημάτων για παράδειγμα, ε, εταιρικέ σχέσεις ανάμεσα σε, σε υπηρεσίες απασχόλησης κλπ. θα αποτελέσουν αντικείμενο αυτής. Τρίτον, ε, συμμετοχική υψηλή ποιότητα, ε, συμμετοχικό ποιότητα διάλογο για την πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον, ε, δημιουργία ε, δικτύων δεξιοτήτων, ε, ανάπτυξη δεξιοτήτων για να προωθήσουμε την ανάπτυξη πολιτικών και στόχων. <clears throat> Θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε τέτοιου δραστηριότητε, παράδειγμα καταπολέμηση των διακρίσεων και πρόθεση των γυναικών στην λήψη αποφάσεων. Τέλο, καλύτερη ενσωμάτωση οριζόντιων θεμάτων, για παράδειγμα ε, προβλήματα τα οποία αφορούν οριζόντια την ισότητα των φύλων, την αποφύγη των διακρίσεων και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ε, το mainstreaming του φύλου, ε, που είναι μία από τις βασικές αρχές, θα εξακολουθήσει να είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του σχεδιασμού και της εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων της πρόοδου. Θα απαιτηθεί συλλογή στοιχείων αναφύλου ε, τέλος, θα ήθελα να σας πω δύο λόγια για ένα πολύ επίκαιρο θέμα που είναι η Λευκή Βίβλος για τις συντάξεις. Το έγγραφο που προετοιμάζουμε <clears throat> θα διαπνέεται από μια ισχυρή ε, ε, προσέγγιση φύλου. Θέλουμε τα συνδεξιωτικά στήματα να είναι βιώσιμα, ε, και επαρκή, μειώνοντα όμω διαφορέ ανάμεσα στι γυναίκε και του άντρε. Η Λευκή Βίβλο θα δημιουργήσει, θέλει να δημιουργήσει τι συνθήκε για μια ισχυρή συμμετοχή και για ανδρών και γυναικών στην αγορά εργασία, μεγαλώντα τον κύκλο ζωή ε, στην, εργασία του και βελτιώνοντα τι ευκαιρίε. Γνωρίζω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανισότητε μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασία. <clears throat> Ανισότητε σε ό,τι αφορά τα ποσοστά συμμετοχή, τι αμοιβέ, ε, τι την καταμερισμό των ευθυνών στην εργασία κλπ. Και αυτά τα προβλήματα, αυτές οι αδυναμίες μπορούν να ε, δυσκολεύσουν τις γυναίκες στο να υποφεληθούν ε, πλήρως της ανεξαρτησίας τους. Αυτές οι δυσκολίες επίσης θα τις ε, δυσκολεύσουν να συμμετάσχουν πλήρως και στην συντάξη τους, <clears throat> οπότε ε, θα, τους, ε, θα τις οδηγήσουν σε χαμηλότερες συντάξεις στο ε, μέλλον όταν μεγαλώσουν. Γι' αυτό λόγο η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει ότι τα θέματα ισότητας των δύο φύλων θα αποτελέσουν ε, αναπόσπαστο τμήμα της Λευκής Βίβλου για τις ε, συντάξεις και τις παρακολούθησής τους. προς, θα υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να μειώσουμε τις διαφορέ διαφορές μεταξύ των δύο φύλων στην αγορά εργασίας και στα συνταξιωτικά συστήματα <clears throat> έτσι ώστε τα μελλοντικά συνταξιωτικά συστήματα να είναι επαρκή, βιώσιμα και ασφαλή για άνδρες και γυναίκες. Ε, θα παρουσιάσουμε την άσπρη βίβλο κατά τη διάρκεια του έτους ε, ενεργής ε, γύρανσης που θα λάβει χώρο το 2012 η ενεργή γύρανση δίνει ευκαιρία σε όλους τους ανθρώπους να κρατήσουν τον έλεγχο της ζωής τους, δίνοντάς τους ευκαιρία ε, να συνεχίσουν να εργάζονται και να τους επιτρέπει να, μέσω εθελοντικής εργασίας ε, να συμμετέχουν στην κοινωνία και να ζουν ανεξάρτητα όσο δυνατό περισσότερο μπορούν. Η Στρατηγική Ευρώπη 2020, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το Πολιετές ε, Δημοσιονομικό Πλαίσιο ε, έχουν συμπεριλάβει παρκή και κατάλληλα μέτρα που μας επιτρέπουν να εκμεταλλευτούμε ε, τις ευκαιρίες ε, σχετικά με το φύλλο που δεν έχουμε ακόμα εκμεταλλευτεί. Συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ελπίζουμε ότι θα καταφέρουμε να εισάγουμε την διάσταση του φύλλου σε όλο και περισσότερες πολιτικές στην ισότητα των να λαμβάνουμε υπόψη το γεγονό ότι οι γυναίκες διαφέρουν από τους άντρες ε, ό,τι αφορά το ρόλο τους στην ιδιωτική ζωή ε, ή, το, το, το ότι είναι περισσότερο ευάλωτες. Ε, η ενσωμάτωση αυτών των χαρακτηριστικών σε διάφορες πτυχές της πολιτικής δεν έχουμε ακόμα εξαλείψει όλα τα εμπόδια στον δρόμο των γυναικών πως ε, οι, οι στόχοι σταθερότητας και ανάπτυξης δεν μπορούν να επιτευχθούν πλήρως. Γι' αυτό το λόγο η ισότητα των δύο φύλων είναι και οικονομική και κοινωνική ανάγκη κατά την άποψή μου. Μην ξεχνάμε ότι για να επιτύχουμε τους στόχους μας πρέπει, χρειαζόμαστε μάλλον, τη βοήθεια των γυναικών αλλά και των ανδρών. Θα πρέπει λοιπόν ο διάλογος να είναι συμμετοχικός, πολυφωνικός και πλήρης για να πετύχουμε και στην απασχόληση και στην κοινωνική ζωή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Με πολύ χαρά μου θα απαντήσω σε ερωτήσεις σας και θα συμμετάσχω στο διάλογο. Ήδη ο πρόεδρος σας είπε ότι έχω κάποιους χρονικούς περιορισμούς. Έχω αναλάβει την δέσμευση να ε, παραστώ και στην συνέντευξη μια άλλη επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά εντωμεταξύ μέχρι τι 4 με πολύ χαρά θα συζητήσω μαζί σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Άντορ, για αυτή την παρουσίαση. Πραγματικά μας πιέζει ο χρόνος, ειδικά εσάς, οπότε, όπως είπαμε και πριν, οι συντονιστές θα έχουν το χρόνο που του δώσαμε, ενώ για του υπόλοιπου συναδέλφου 1,5 ή 1 λεπτό μόνο έχουν στη θέση του για να μπορέσει να έχει το χρόνο ε, και ο να απαντήσει. Κύριε Σπαλά. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Oh, sorry. Yeah, I say that uh, if you wanted... Ζητώ συγγνώμη αν δεν ακούσετε τη διερμήνεια. Σα έδωσα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Η ισότητα των φύλων είναι ένα θέμα αρμοδιότητας δύο επιτρόπων. Αυτό, παρά τα αυτά, δίνει όλο και λιγότερο χρόνο και χώρο για τις δύο θεμάτων. Οπότε λαμβάνουμε τις πυρήνες παρουσίας ως χριστουγεννιάτικο δώρο στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε θερμά λοιπόν για την παρουσία σας. Θα ήθελα να θέσω μία σειρά ερωτημάτων, μου επιτρέπετε. Αναφερθήκατε στρατηγική του 2020 και τις όλες ανησυχίες γύρω από το θέμα μας απασχολεί. Να πω ποιες είναι οι δικές μας ανησυχίες. Ακόμα και αν η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη παρά τις προσπάθειες που κάνουν δεν καταβάλουν πραγματικά απ βήματα για να επιτύχουν το 75% τη απασχολησιμότητα των γυναικών. Αυτός ο στόχος δεν πρόκειται να επιτευχθεί από μόνος του. Θεωρώ ότι είναι ε, προφανές για όλους αυτό. Δεν έχει νόημα καν, πιστεύω, να μιλούμε για τους στόχους Βαρκελόνη. διότι ε, οι κυβερνήσεις δεν αρέσκονται να μιλούν γι' αυτό. Έχω όμω την αίσθηση ότι το να ξεχνούμε τους στόχους Βαρκελόνης είναι πρόβλημα. Όταν μιλούμε για στρατηγική 2020 και μιλούμε συγκεκριμένα για την ελάφρυνση και τη μείωση της φτώχειας, Έχω την αίσθηση ότι πολλέ φορέ μιλούμε για διαφορετικά πράγματα, διαφορετικούς στόχους. Έχουμε δημιουργήσει κάποιου στόχους ενώ τη 2020, αλλά η πραγματικότητα έχει αλλάξει στο μεσοδιάστημα. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε 20 εκατομμύρια παιδιά κάτω από το όριο της φτώχειας. Και υπάρχουν και άλλα στατιστικά στοιχεία που ακόμη δεν τα γνωρίζουμε. Ρωτώ, τι θα κάνουμε γι' αυτό. Και ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί βλέπω ότι ο πρόεδρος ε, με κοιτά αρκετά έντονα. Όσον αφορά τη γύρανση, δεν έχουμε στατιστικά δεδομένα, δεν ξέρουμε πώς έχει αυτή την κατάσταση, όμως είναι προφανές ότι οι γυναίκες γυράσκουν διαφορετικά από τους άνδρες είναι πολύ μεγαλύτερο το βάρος που φέρουν οι γυναίκες ε, ε, καθώς περνούν τα χρόνια. Ε, τι προτίθεστε να κάνετε για αυτό το ζήτημα, τι θα κάνετε ακριβώς για να προσπαθήσετε καλύτερα τις γυράσκουσες γυναίκες. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος δύο λεπτά. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επιτρόπε, δύο ερωτήματα. Πρώτα απ' όλα για το mainstreaming των ε, φίλων και πώς συνδέεται αυτό με τα διευθυντικά ταμεία. Από ό,τι βλέπω από τη δική μου χώρα, από τη Δανία, είναι ότι καμία ε, δεν θα λέγαω ότι δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη η διάσταση του φύλου α, από κανένα διευθυντικό ταμείο, ούτε περιφερειακό, ούτε κοινωνικό ταμείο. Πουθενά, πουθενά στην ταμείο δεν έχω ακούσει τη λέξη gender mainstreaming. Και αυτό με ανησυχεί διπλά. Γιατί προς το παρόν, αυτή τη στιγμή, έχουμε στο τραπέζι μια νέα οδηγία με στόχο τη δημιουργία περισσότερων οικολογικών εργασία. Και μάλιστα η νέα Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα τους ορμητοφορείς και ε, μια άλλη προτεραιότητα είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας σε αυτό τον τομέα. Μήπως όταν μιλούμε για αυτές τις οικολογικές εργασίες θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διάσταση των γυναικών πουθενά δεν γίνεται ειδική αναφορά για τις γυναίκες και την απασχόληση. Πιστεύω ότι η Επιτροπή πρέπει να κάνει κάτι εν προκειμένου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί και πάντοτε όταν συζητούμε για τη δημιουργία πράσινων οικολογικών θέσεων εργασία, πάντοτε αναλαμβάνουμε υπόψη και τη διάσταση των γυναικών στα πλαίσια γενικότερα τη συνεκτίμηση διάσταση του φύλου στι πολιτικέ. Δεύτερο ερώτημα είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω μία αποστολή για τους Ρωμά. Και ειδικά το θέμα των γυναικών ήταν κάτι που μας απασχόλησε. Κατά τη διάρκεια της Ουγγρικής Προεδρίας Είχαμε θέσει στο τραπέζι το θέμα των Ρωμά ω μια στήρευτη πηγή εργασία. Τι γίνεται με τι γυναίκε Ρωμά εν προκειμένου, την ένταξή του στην κοινωνία και πώ προωθεί τη χρηματοδότηση και η ενίσχυση αυτών των ομάδων πληθυσμού. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπάντον, δεν είναι εδώ. Θα ήθελε κανείς από το άλλο το λόγο. Όχι. Η κυρία έχει ένα λεπτό και 30 διάθεσή uh, ε, Ευχαριστούμε πολύ για την έλευσή σας κύριε Άντορ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Στη Επιτροπή Απασχόλησης, ε, στη... μάλλον είμαι ε, υπεύθυνη για την έκθεση στην Επιτροπή Απασχόλησης. Μιλούμε για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και το ε, πρόγραμμα για το 2020. Ε, μιλούμε για τις απεριόριστες δυνατότητες ε, που έχουν οι γυναίκες και θεωρητικά θα έλεγα ότι είναι θαυμάσιο να έχουμε αυτούς τους στόχους του 2020, τους οικονομικούς, τους κοινωνικούς ε, και το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο μας φέρνει πιο κοντά σε όλα αυτά. Αλλά στην πράξη τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται ότι είχαμε τα αποτελέσματα τα οποία ελπίζαμε. Ε, παντού μένεται ένας αγώνας αρμοδιοτήτων στο Συμβούλιο, στην, στο ΕΚΟΦΗΝ, στην, ε, στο Συμβούλιο Απασχόλησης, ενώ εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε την Επιτροπή Απασχόλησης, αφενός την Επιτροπή Γυναικών αφετέρου και επίσης και η Γενική Διεύθυνση ε, Περιβάλλοντος και η Γενική Διεύθυνση ε, Κοινωνικών Υποθέσεων Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ε, αντιμάχονται η μία την άλλη για τα 15 αυτά εκατομμύρια 215 εκατομμύρια των γυναικών Επίσης δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα της ισότητας, ισότητας των φύλων ε, ε, στην τελευταία έκθεση και θα ήθελα να μάθω τι θα γίνει για να περιληφθεί και η διάσταση της ενσωμάτωσης των δύο φύλων στις, στα νέα προγράμματα και τις ε, μεταρρυθμίσεις. Ενώ θέλω να μάθω στην έκθεση ε, Μπρέστα εμείς ζητήσαμε να υπάρξει μια σκιώδης έκθεση σχετικά με τις ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα γυναικών. Ευχαριστώ, Επιτροπέ. Είναι ενδιαφέρουσα η περίοδος που ζούμε και ασφαλώς το θέμα της απασχόλησης θα παίξει κρίσιμο ρόλο στην ανάπτυξη. Οι γυναίκες καταρχήν έχουν μια επιλογή να δουλέψουν ή να μην δουλέψουν και ό,τι και αν πράξουν είναι πολύτιμο. Και με ενδιαφέρον παρακολούθησα το σχόλιο σας για τις διαφορές που αναγνωρίζονται και για τη δράση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Όπως γνωρίζετε, ε, είμαι κατά της άδειας ε, μητρότητας. Όχι επειδή είμαι κατά της έννοιας, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ε, και άλλοι τρόποι για να βοηθήσουμε τις γυναίκες στην απασχόληση. Και υπάρχει και η δυνατότητα της άδεια του πατέρα. Είναι λιγότερο περιγραφική και επιτρέπει λιγότερες διακρίσεις. Είμαι λοιπόν υποστηρικτής αυτής της ιδέας και με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται οι ανάγκες της οικογένειας. Ε, ε ποια είναι λοιπόν η άποψή σας σε σχέση με αυτό και σε συνδυασμό με την άδεια μητρότητας. Τώρα, Υπάρχει το άλλο θέμα των ποσοστώσεων. Ποια είναι η άποψή σα, Οι γυναίκε μπορούν να καταφέρουν, τα καταφέρουν μόνε του ή χρειάζεται μια όθηση. Και ένα τελευταίο στοιχείο σχετικά με τι συντάξεις. Ναι, πράγματι θα πρέπει να συνδέονται με τη διάσταση του φίλου και έχουμε την περίπτωση ε, την πρόσφατη περίπτωση και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια αξιολόγηση των κινδύνων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι το θέμα των συντάξεων θα πρέπει να ανήκει στην αρμοδιότητα των κρατών. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Φιγκουρέντο δεν είναι εδώ. Η κυρία Σανκλέρ για ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της, του φίλου ε, στην λήψη αποφάσεων πιο συγκεκριμένα. Και εγώ διαφωνώ με τις ποσοστώσεις, όπως είπε και η κυρία Γιανακουδάκη. Ε, δημιουργούν σημαντικά προβλήματα ιδιαίτερα στι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και συνεπώς σε όλη την οικονομία και την απασχόληση. Πιστεύετε όμως ότι δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υλοποιεί αυτά που κηρύττει. Μόνο εννέα είναι οι γυναίκες επίτροποι. Ε, ο στις 22 προέδρους επιτροπών στο Κοινοβούλιο είναι γυναίκες. Ε, το ψηλότερο ποσοστό νομίζω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, αν η Κομισιόν από μόνη τη δεν προωθεί αρκετά τι γυναίκε, γιατί πιστεύετε ότι οι μικρομισέ επιχειρήσει ή επιχειρήσει γενικότερα ε, θα δώσουν περισσότερο λόγο στις γυναίκες. Ε, εδώ πέρα έχουν προβλήματα και με την ομοθεσία. Πολύ δε περισσότερο με τι ποσοστώσει. Ε, θα Πρέπει να υλοποιούμε αυτό που κηρύττουμε, να το θέτουμε σε πράξη. Πρόεδρος. Uh, euh, ε, ευχαριστώ, Επίτροπε, που είστε μαζί μας. Ε, πρώτο σχόλιο, σε ό,τι αφορά τους μισθούς. Είπατε ότι πολύ συχνά ο μισθός γυναίκας είναι δεύτερο εισόδημα για τον οικοκυριό. Πώς θα μπορούσαμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να αναθεωρήσουν το φορολογικό του σύστημα έτσι ώστε ο μισθός των γυναικών να μην είναι πρόσθετος έναντι του μισθού του άντρα αλλά να είσαι ε, ίσος, ισότιμος. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την καριέρα Εκεί πρέπει να κάνουμε σημαντική προσπάθεια γιατί σήμερα όσο γεννιόνται παιδιά σε μια οικογένεια η γυναίκα εργάζεται όλο και λιγότερο. Οπότε τα κράτη και οι οικογένειες επενδύουν όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση των κοριτσιών οπότε γιατί δεν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις γυναίκες όταν μεγαλώσουν στην καριέρα τους. Τρίτον, ε, ε, έχουμε θέσει όρους σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση από το Κοινωνικό Ταμείο ε, και οι όροι αυτοί ως τώρα ε, αφορούσαν τη χρηστή διαχείριση. Γιατί δεν βάζουμε και ένα πρόσθετο όρο για την εισαγωγή του, της πτυχής του φύλου στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Κοινωνικό Ταμείο. Μετά, ζητούμε, απαιτούμε πολλές προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πλάν. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την παρουσία σα εδώ. Θεωρούμε ότι είναι ένα κομβικό ρόλο, ειδικά αυτή την περίοδο κρίσης. Είπατε ότι είναι κοινωνική και οικονομική ανάγκη η ισότητα των φύλων και καλείται τα κράτη-μέλη να προωθούν την ισότητα των φύλων με την συνεκτίμηση διάσταση του φίλου στι πολιτικές και ειδικέ Και ρωτώ, αν τα κράτη-μέλη δεν σεβαστούν τις δικές σας εκκλήσει, τι θα γίνει. Μπορείτε να παρέμβετε στα εσωτερικά των κρατών μελών. Μπορώ να σας πολλά παραδείγματα. Γνωρίζετε πολύ καλά και εσείς ο ίδιος ότι θέλετε να κάνετε πολύ καλή δουλειά στο θέμα της ε, διάστασης του φίλου Ρωτώ, μπορείτε, μπορείτε να παρέμβετε στα ιστορικά των κρατών μελών αν δεν σεβαστούν αυτές οι εκκλήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλος το λόγο να θέσει ερωτήσεις, οπότε θα δώσω το λόγο στον Επίτροπο να απαντήσει στα ερωτήματα. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετό χρόνο μέχρι να πρέπει να μα εγκαταλείψετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα και σχόλια. Κάποιε φορέ τίθεται ερωτήματα, αλλά είναι πιο πολύ σχόλια παρά ερωτήματα. Το βασικό θέμα που ήρθε και επανήλθε σε πολλές παρεμβάσεις είναι το θέμα των στόχων. Κατά πόσο οι στόχοι της Ευρώπης 2020 σχετικά με την επασχόληση και τη φτώχεια, κατά πόσον είναι οι γενικότεροι στόχοι που περιέχουν τη διάσταση του φύλου ή πρέπει να έχουν πιο ειδικούς στόχους. Και αυτό αφορά την αναλογικότητα των γυναικών σε ηγετικέ θέσει εργασία. Οι στόχοι έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να υπάρξει συμφωνία επί των στόχων και να θέσουν, αν θέλετε, ένα πεδίο εφικτό για να επιτύχουμε την ανάπτυξη. Αν όμω είναι μη ρεαλιστική η στόχη, τότε δεν υπάρχει και κανένα κίνητρο για να επιτευχθούν οι στόχοι και άρα να συμμετέχουν όλο και περισσότεροι φορείς. Να ξεκινήσω από το πρώτο. Κατά πόσο το 75% ο στόχος είναι ρεαλιστικός στόχος. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αντίθετες προβλέψεις. Αν λοιπόν υπάρξει μια κρίση μάζα πολιτικών, μπορούμε να το επιτύχουμε, αλλά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι πολύ αρνητικά και δεν βλέπω να μπορούμε με τις υφιστάμενες πολιτικές να επιτύχουμε αυτό το στόχο. Αλλά θα είμαι και ειλικρινής. Όταν ορίστηκε ο στόχος του 75% πριν από 18 μήνες περίπου και υιοθέτησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό έγινε μετά την τόσο παρτεταμένη οικονομική κρίση που βιώνουμε σήμερα και που φοβούμε ότι δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Αντί λοιπόν όλα αυτά να βοηθούν την ανάπτυξη απασχόλησης, το αντίθετο βλέπουμε να συμβαίνει, βλέπουμε να συνεχίζει η ύφεση και μείωση των ποσοστών απασχόλησης στον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Αυτή είναι η εικόνα της παρούσης κατάστασης και άρα η συγκυρία δεν μας επιτρέπει να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Ίσως κάποια στιγμή να απαιτηθεί να αναθεωρήσουμε αυτούς τους στόχους. Όμως αυτή τη στιγμή είμαστε στις πρώτες φάσεις στρατηγικής 2020. Αυτό που εγώ προσπαθώ να υποστηρίξω είναι ότι οι πολιτικές θα πρέπει να αναθεωρούνται και να ενισχύονται και να αυξάνονται οι προσπάθειες. Όχι να μειώνουμε, αν θέλετε, τον πύχη των προσδοκιών. Αυτό θα κάνουμε ε, ήδη το 2012 με ένα νέο πακέτο, με μια ευρεία δέσμη πολιτικών και η διάσταση του φύλου είναι κομμάτι αυτού του πακέτου, του κοινωνικού πακέτου που ετοιμάζουμε για την επόμενη χρονιά. Κυρία Παύλη μίλησε για τους στόχους της στόχες. Ναι, είναι τόσο μεγάλο ο αριθμό των θέσεων εργασία που ε, χάνονται και λόγω της δημοσιονομικής εξυγίανση, η κατάσταση είναι δύσκολη κατά μέσο όρο. Και αυτό που είναι πιο προβληματικό είναι ότι η Ευρώπη είναι όλο και πιο δικασμένη από ποτέ. Υπάρχει και μεγάλη ασυμμετρία, περισσότερο από ποτέ, και αυτό σημαίνει ότι στις ε, περιφερειακές, αν θέλετε, χώρες της Ευρώπης, το λέμε έτσι απλουστευτικά, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Σε ό,τι αφορά τους στόχους, όπως ε, ε το 1 τέταρτο ε, για τα θέματα του φίλου, νομίζω ότι είναι στόχοι που έχουν ορθά επιλεγεί. Και οι καταληκτικές προθεσμίες είναι εφικτές. Έχουν νόημα αυτοί οι στόχοι. Πιστεύω ότι οι στόχοι δεν θα πρέπει να είναι τόσο ποσοτικοί, θα έλεγα, σε αυτό το τομέα πολιτική Το έχω συζητήσει αυτό το θέμα πολλές φορές και με τον και συμμεριζόμαστε την ίδια θέση, θα έλεγα. Αν σε αυτό το τομέα τελικά δεν αποβούν αποτελεσματικά ήπια εργαλεία, εργαλεία ήπιας ε, ε, πολιτικής, ίσως θα πρέπει να δούμε το θέμα αν θέλετε διαφορετικά. Επίσης, οι, στόχοι και οι ποσοστώσεις δεν θεωρώ ότι λειτουργούν ματροναριστικά. Ε, η κοινότητα πολιτών εν και οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να βοηθήσουν σε αυτήν την κατεύθυνση για να επιτύχουμε αυτό τον στόχο που ασπαζόμαστε όλοι. Τώρα, κατά πόσο αυστηροί μπορούμε να είμαστε σχετικά με τους στόχους που θέσαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξαρτάται από το εκάστοτε ζήτημα. Όσον αφορά τι συστάσει που απευθύνουμε σε κάθε χώρο διαφορετική, όπω είναι η δημιουργία εγκαταστάσεων για τη φροντίδα του παιδιού, είναι κάτι που ήδη υπάρχει σε επιμέρους συστάσεις, όπως και η εξίσωση των ε, ηλικιακών ορίων σταξιοδότηση μεταξύ ανδρών και γυναικών. Είναι ένα ισχυρό εργαλείο αυτό. Σε άλλου τομεί όμω, όπου νομικώ πώ η αρμοδιότητα είναι εθνική, εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω άλλων παρεμβάσεων, μέσω άλλων μέτρων, πιο πολύ υποστηρικτικών μέτρων, μπορεί να διαδραματίσει ισχυρό ρόλο και να καταφθύνει, αν θέλετε, ε, τις εξελίξεις. Είναι πάντως πολύ σημαντικό να υπάρξει πολιτική βούληση και πολιτική δέσμευση. Αν δεν υπάρξει δέσμευση, βούληση πολιτική σε τοπικό εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι όσο αυστηρή θέλει και να κάνει αν θέλετε, τον ε, αυστηρό δάσκαλο. Αλλά πιο σημαντικό είναι να υπάρξει συνειδητοποίηση και γρήγορση σε τοπικό επίπεδο. Εμείς στηρίζουμε τη δράση κοινωνίας των πολιτών, εκστρατείες ενημέρωσης, πιλωτικά προγράμματα που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε καλές πρακτικές και να τις διαδώσουμε περαιτέρω. Και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο τα κράτη-μέλη μπορούν να χρηματοδοτήσουν προγράμματα που θα έχουν πολλαπλασιαστικό, αν θέλετε, αποτέλεσμα. Σχετικά τώρα με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο που εισέρχεται στην δεύτερη φάση. Ανέφερα ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συστάσεις ανάλογα με τις χώρες και αυτό είναι ένα ισχυρό μέσο, εργαλείο και συμφωνώ ότι αυτό είναι και απολύτως νόμιμο. Αν δηλαδή οι στόχοι και οι συστάσεις αναπτυχθούν με έναν ισόρροπο τρόπο. Και το δικό μου χαρτοφυλάκιο διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο. Στο πρώτο εξάμεινο υποβάλαμε τα τεκμήρια σε συνεργασία με την ΕΚΦΗΝ. Τώρα ε, εισέρχεται και το θέμα της φορολογίας, διότι θέλουμε ισότητα και στις, ε, στην χρηματοδότηση και στην ένταξη στην αγορά και στα δημόσια οικονομικά. Είναι ε, ένα επίγον θέμα που θα συμβάλλει στην ορθή οικονομική ανάπτυξη. Όταν υπάρχει οικονομική αστάθεια, βεβαίως τα βραχυπρόθεσμα μέτρα είναι αυτά που κυριαρχούν. Από τη στιγμή λοιπόν που η Ευρώπη θα ξεπεράσει αυτά τα βραχυπρόθεσμα ε, προβλήματα, θα είναι πολύ πιο εύκολο να προχωρήσει σε μια πιο ισόρροπη πολιτική. Ε, διαφορετικά το κόστος αυτής της ύφεσης θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Στο μέτρο του δυνατού πιστεύω ότι πράττουμε αυτό το οποίο διδάσκουμε, διακηρύττουμε και αναπτύσσεται ένα σχήμα απασχόλησης ορθό υποστηρίζονται πολιτικές που ενθαρρύνουν την συμμετοχή και την ισόρροπη συμμετοχή των δύο φύλων και σε πολιτικές θέσεις αλλά σαφώς πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά στον τομέα αυτό. Το να δίδουμε το σωστό παράδειγμα πάντα βοηθάει. Εγώ είμαι ίσως ο μόνος επίτροπος που έχει επικεφαλής του γραφείου αλλά και αναπληρωτή γυναίκα. Και επειδή ομιλώ στο σωστό ακροατήριο, πραγματικά θέλω να δώσω το παράδειγμα. Αλλά όταν καλείς επιβάλλει αυστηρούς όρους και ποσοστώσεις ε, και λοιπά, σίγουρα αυτό θα προκαλέσει διαμαρτυρίες. Άρα λοιπόν θα πρέπει κανείς να αναζητήσει μια ισορροπία, δηλαδή να συνδυάσει τα ισχυρά εργαλεία, αλλά επίσης και να αναπτύξει τα κατάλληλα πολιτικά επιχειρήματα και να πείσει τους ε, ε, πολίτες για έναν πολύ ορθό στόχο. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό. Ο Πρόεδρος, Ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε αφιερώσει τον χρόνο να έρθετε στην Επιτροπή μας. Έτσι μπορέσαμε να έχουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων μαζί σας. Ε, όπως είπα και στην αρχή, εδώ και καιρό θα θέλαμε να σας έχουμε μαζί μας και τελικά το καταφέραμε. Ήταν πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή απόψεων, κάτι το οποίο θέλουμε να συμβαίνει συχνά. Ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά. Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε λοιπόν. Όπως είπα και προηγουμένως, περνούμε τώρα στο σημείο 7 της ημερησία διάταξης απασχόληση και κοινωνικές πτυχές στην ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2012. Και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κορνίλσεν ευθύς αμέσως. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι λογικό να ασχοληθούμε με το σημείο αυτό αμέσως μετά την παρέμβαση του κυρίου Άντορ, διότι ήδη συζητήσαμε μαζί του το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είμαι η συγγήτρια στην απασχόληση και θα κάνουμε και τροπολογίες στην έκθεση αυτή. Ελέγχθησαν πολλά για την σημασία της διάστασης των φύλων το πρόγραμμα Ευρώπη 2020 και το εξάμεινο. Εμείς λοιπόν ως Κοινοβούλιο νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ισχυρή θέση. Ε, δεν λέει πουθενά το κείμενο ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες, άρα έχουμε αρμοδιότητες και έχουμε ψηφίσει και τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου που μπορούμε να στείλουμε στο Συμβούλιο ώστε να ληφθεί η υπόψη στη διάσκεψη κορυφής της ε, Άνοιξης και ελπίζει κανείς ότι θα φτάσουμε κάπου. Εγώ στην έκθεσή μου εντοπίζω πέντε προτεραιότητες. Θα προσπαθήσω να πείσω το Κοινοβούλιο να δεχθεί τις προτεραιότητες αυτές αντί να βάλουμε όλα τα θέματα στο ίδιο καλάθι. Πολλά από τα θέματα αυτά συνδέονται με το ζήτημα της ισότητας των φύλων διότι οι φιλοδοξίες φοβούμε ότι είναι πολύ χαμηλές σε πάρα πολλά μεταρρυθμιστικά προγράμματα των χωρών το θέμα της ισότητας δεν αναφέρεται καν. Έχετε λοιπόν τις προτάσεις μου σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων. Αύριο είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών στην Επιτροπή Απασχόλησης. Αν υπάρχουν άλλες προτάσεις, ε, άλλες τροπολογίες για την έκθεση αυτή, με μεγάλη χαρά θα τις περιλάβω, αν βεβαίως συμφωνώ με αυτές. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Έχετε το λόγο στο θέμα αυτό. Έχετε το λόγο. Ποιος θα ήθελε να λάβει το λόγο, παρακαλώ. Thank you so much. Thank you. Ευχαριστώ για την ευκαιρία αυτή και ευχαριστώ για τις ενδιαφέρουσες και ολοκληρωμένες τροπολογίες. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις για να κατανοήσω καλύτερα τις αρχικές προθέσεις. Στην τροπολογία 7. Θα ήταν καλό να γνωρίζουμε τι επιδίωκε ο συντάκτης όταν μιλάει για αυτόματους κοινωνικούς σταθεροποιητές. Αντιλαμβάνομαι ότι μιλάει για το σύστημα κοινωνικής προστασίας, αλλά ποιοι είναι αυτοί οι αυτόματοι κοινωνικοί σταθεροποιητές, δεν είναι απόλυτα σαφές για μένα. Υπάρχει ακόμα ένα θέμα όσον αφορά την τροπολογία υπαριθμών εννέα. δεν είναι απόλυτα σαφές τι ζητούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει δηλαδή να γίνει μια ανάλυση ε, μια ανάλυση της ε, επιρροής της διάστασης ε, της ενσωμάτωσης της ισότητας των δύο φύλων στις μεταρρυθμίσεις των ε, συνταξιδοτικών προγραμμάτων ε, και αυτό βεβαίως ω συνέπεια στη ζωή των γυναικών. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς περί πρόκειται. Ο Πρόεδρος. κυρία Κορνέλσεν θα θέλατε να εξηγήσετε. Ίσως μπορούμε να το επαναδιατυπώσουμε αν δεν είναι αρκετά σαφές. Αυτόματοι κοινωνικοί σταθεροποιητές. Συνήθως η κοινωνική ασφάλιση λειτουργεί ως αυτόματος σταθεροποιητής για να διατηρηθεί η αγοραστική αξία ας πούμε ε, με το ύψος της ε, ε, σύνταξης. Ε, ή της αμοιβή. Δηλαδή, όταν κανείς χάνει τη δουλειά του δεν μπορεί να αγοράσει αυτά τα οποία ε, θα μπορούσε να αγοράσει. Υπησέρχεται λοιπόν το κοινωνικό σύστημα ως σταθεροποιητής. Θα μπορούσαμε όμως να επαναδιατυπώσουμε την τροπολογία για να γίνει πιο σαφής. Τροπολογία υπαριθμών 9. Η έρευνα ετήσιας ανάπτυξης προτείνει να ληφθούν μέτρα ώστε οι συντάξεις να είναι εφικτές οικονομικά στο μέλλον. Εδώ αναφέρονται συγκεκριμένα οι συντάξεις, διότι πράγματι πρόκειται για το μεγαλύτερο έξοδο που έχουν να καταβάλουν οι κυβερνήσεις. Και τώρα σχεδόν όλες οι χώρες ε, προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις των συνταξιδοτικών του συστημάτων. Άρα λοιπόν και αυτό θα πρέπει να ειδωθεί και να το προσεγγίσουμε και από τη σκοπιά της ισότητας των δύο φύλων. Μεταρρυθμίσεις, τις μεταρρυθμίσεις λοιπόν αυτές να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να συνδυαστεί με άλλα μέτρα ως προς το εισόδημα και την φορολογία. Διότι μερικές φορές τα μέτρα που λαμβάνονται για τις συντάξεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα μέτρα που λαμβάνονται ε, σε φορολογικό επίπεδο. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση για να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις συγκεκριμένα στο εισόδημα των γυναικών μετά από όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν η Κομισιόν θα ήθελε να πει κάτι. Κομισιόν, θέλει το λόγο. Όχι. Και κανείς άλλος κιόλας. Ωραία. Αφήνουμε πίσω μας λοιπόν αυτό το θέμα και περνάμε στο 15 όπως είχα ανακοινώσει. όπως είπε η κυρία Κορνέλησεν, θα ψηφιστεί το, η έκθεση της αύριο. Ε, αυτό το ξέχασα να σας το πω, το είχε δει η κυρία Κορνέλησεν. Ωραία. Έχοντας κλείσει και αυτό, περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν, όπως είπα. 15 Σημείο 15 όπως είπα. Μισό δευτερόλεπτο να βρω τα χαρτιά μου. Ε, ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2011. Αυτός είναι ο τίτλος. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Ιντβέλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ζητώ συγγνώμη από τους συναδέλφους. Σας είχα πει από την αρχή ότι θα πρέπει να φύγω σε 10 λεπτά, 15, γιατί πρέπει να συναντηθώ με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, δύο λόγια λοιπόν να σας πω. Πρόκειται για την ετήσια έκθεση ισότητας μεταξύ άνδρων και γυναικών. Ως γενική παρατήρηση να πω το εξή. Ας σκεφτούμε λίγο περισσότερο το πώς θα επηρεάσουμε περισσότερο τα πράγματα της πολιτικής ισότητας ήδη νωρίτερα σήμερα στην ανταλλαγή απόψεων με τον Επιτροπή και ο Άντορ είπαμε ότι εμείς μπορεί να υιοθετούμε και να εγκρίνουμε όλους αυτούς τους πολύ ε, καλούς στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά το θέμα είναι να υλοποιούνται και από τα κράτη-μέλη, γιατί αλλιώς οι αιτήσει εκθέσεις ε, γίνονται απλώ μια ε, ρουτίνα. Κατά τα άλλα, τα εξής βασικά σχόλια. Οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Πολλέ παρατηρήσεις για τα θέματα αυτά έχουν ήδη γίνει τα προηγούμενα χρόνια, οπότε δεν θέλω να επαναλαμβάνω τα πάντα. Έτσι. Ε, απλώς ε, εστιάζω στα καινούρια. Πρώτον, μία αναφορά στην ε, διαφορά αμοιβή μεταξύ άντρων και γυναικών που επιμένει ε, παρόλο ότι προσπαθούμε να τη μειώσουμε, δεν έχουμε σημαντικά αποτελέσματα, χρειαζόμαστε ένα οδικό χάρτη. Εν παρενθέσει, να πούμε ότι ε, παρόλο ότι εστιάζουμε στην ενίσχυση του ρόλου της γυναίκας στην αγορά εργασίας, ίσως θα έπρεπε να δούμε και το μέλλον και να διαπιστώσουμε ότι τα κορίτσια και τα, ε, οι νέες γυναίκες ξεπερνούν σε επιδόσεις τα αγόρια και τους νέους άντρες. Οπότε στο μέλλον, δεδομένου ότι η οικονομία είναι όλο και περισσότερο μια οικονομία υπηρεσιών και γνώσης, αυτοί που θα έχουν λάβει την καλύτερη εκπαίδευση θα είναι σε καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους. Συνεπώς, ενδεχομένως, η κατάσταση μεταξύ άντρων και γυναικών μπορεί να αντιστραφεί μόνο και μόνο εξαιτία αυτών των επιδόσεων των γυναικών που είναι ανώτερες από των αγοριών. Κάνω μια δεύτερη αναφορά σε κάτι το οποίο γνωρούμε πολύ συχνά. Μιλούμε για τα στεξιωτικά δικαιώματα των γυναικών και την ανισότητα στην αμοιβία, αλλά πολλές φορές ξεχνάμε την ε, σε επιπτώσεις του οικογενειακού δικαίου στην οικονομική κατάσταση των γυναικών. Οι στατιστικές στη χώρα μου, ας πούμε, δείχνουν ότι οι γυναίκες μετά από ένα διαζύγιο χάνουν περίπου το 25% του εισοδήματός τους, ενώ οι άντρες κερδίζουν 7%. Θα πρέπει και αυτό λοιπόν να το εντάξουμε στο πλαίσιο της συζήτησης της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών. Μετά, λέω μερικά πράγματα για τις ποσοστώσεις που εν γέννη δεν μας βρίσκουν σύμφωνους, ανα, παραπέμπω σε παλιότερες εκθέσεις. Θα ήταν πολύ χρήσιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταγράψει τα όσα έχουν υιοθετήσει τα κράτη-μέλη και τα αποτελέσματά τους. Μετά ο δεύτερος άξονας, ισότητα των, μεταξύ των κοινωνικών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δηλαδή η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην εξωτερική μας πολιτική ε, όλοι γνωρίζουν την διάσταση του φίλου στην Αραβική Άνοιξη οπότε θα έπρεπε να ενθαρρύνουμε την είπατε εκπρόσωπο και γενικότερα την Κομισιόν να αποδώσουν ιδιαίτερη σημασία σε αυτή την πτυχή γιατί χώρες ε, του αραβικού κόσμου μπορεί να κέρδισαν την δημοκρατία και την ελευθερία, αλλά ενδεχομένως οι γυναίκες ε, να μην κερδίσουν τίποτα και ίσως και να χάσουν κιόλα. Δεύτερο θέμα σε αυτό το κεφάλαιο, η πολύ ανησυχητική εξέλιξη, η μη εξέλιξη για την ακρίβεια, του στόχου της χιλιετίας παρθών 5. Βελτίωση δηλαδή της υγείας των γυναικών, των μητέρων. Ε, στόχο τον οποίο στερούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο εξαιτία ε, έλλειψη χρηματοδότηση. Ε, ο στόχο αυτός έχει σχέση με την αλλαγή νοοτροπία. ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών. Σημαντικό, ε, σημαντικό εμπόδιο λοιπόν αυτό στην επίτευξη του στόχου υπερθών 5, των στόχων της χιλιετίας. Τρίτο ζήτημα σε αυτό το κεφάλαιο αυτό το οποίο ε, ονομάζω αξιοπρέπεια και σωματική κυριότητα των γυναικών ε, ε, βία εναντίον των γυναικών, ομοφιλοφοβία. Η οικιακή βία πολλές φορές θεωρείται ιδιωτικό ζήτημα, εσωτερικό ζήτημα των οικογενειών. Ε, η Ισπανική Προεδρία καλώ το ανέδειξε. Πρόκειται για ένα κοινωνικό ζήτημα. Κοιτάξτε τον τεράστιο αριθμό θυμάτων και θα πιστείτε. Ίσως βέβαια υπερβάλλω λιγάκι λέγοντας ότι θα πρέπει να θεωρηθεί ως θέμα δημοσίας τάξεως ε, αλλά σίγουρα χρειάζεται πολύ περισσότερη προσοχή από ό,τι του αποδίδουμε σήμερα. Μετά αναφέρομαι και πάλι στην σημασία των ε, αναπολιτικών ε, δικαιωμάτων συνδεμένων με τα θρησκευτικά δικαιώματα. Γνωρίζω ότι για κάποιους αυτό είναι ταμπού, αλλά όταν θέλουμε να προστατεύσουμε τις γυναίκες από την ε, σεξουαλική βία, την οικογενειακή βία, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτές τις πτυχές. Τέλος, τρεις παρατηρήσεις που θέλω να συμπεριλάβω. Πρώτον, ελπίζω ότι η δανική προεδρία, η μελλοντική δανική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, θα κάνει πρόοδο στην οριζόντια οδηγία, εναντίον των, το πακέτο δηλαδή εναντίον των διακρίσεων. Δεύτερον, κάνω μια αναφορά στα νοικοκυριά, ε, τα μονογονεϊκά νοικοκυριά, ε, πολύ συχνά δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στις οικογένειες, ε, ε τις πλήρες οικογένειες, αλλά μην αγνοούμε ε, τα δημογραφικά στοιχεία. Ένα στα τρία νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά μέσο όρο είναι μονογονεϊκό. Αυτό δημιουργεί σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση, τη στέγη, την ασφάλεια, τα στεξιδοτικά δικαιώματα, τις κοινωνικές παροχές κλπ. Πρόκειται για ένα στα τρία νοικοκυριά. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Είναι μια εξέλιξη που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος, να επαναλάβω την έκκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει ένα, τελικά επιτέλους ένα, χάρτη, ένα οδικό χάρτη για την ισότητα για τα άτομα της κατηγορίας ΛΟΑΤ, λεσβίες, ομοφιλόφιλοι, αμφιφιλόφιλοι και τρανσεξουαλικοί. Υπάρχει ένα οδικό χάρτη για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Χρειάζεται λοιπόν και ένα παρόμοιο χάρτη για τα άτομα ΛΟΑΤ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Α ξεκινήσει ο διάλογο. Κύριε Τόμψον. Ευχαριστούμε για την εκθεσή σα, κύριε Ενφέλτ. Είναι πολύ καλή. Νομίζω ότι αναδεικνύεται πολύ σημαντικά ζητήματα. Θα μπορούσαμε να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες για την οικιακή βία ή την ε, βία με βάση το φύλλο. Γιατί είναι πραγματικά ε, ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ε, εγώ πράγματι θεωρώ ότι πρόκειται για δημόσιο και όχι για ιδιωτικό ενδοοικογενειακό πρόβλημα. Ας μην ξεχνάμε ότι όλο και περισσότερε γυναίκες στην Ευρώπη πεθαίνουν εξαιτία τη ενδοοικογενειακή βία και πιο πολλέ από ότι ε, ε, αυτές που πεθαίνουν εξαιτία τρομοκρατικών δράσεων. Πλην όμως ε, καταπολεμούμε την τρομοκρατία με πολύ περισσότερα κονδύλια. Επίσης, ε, θα ήθελα να κάνουμε μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Προστασία. και να επιμείνουμε ε, για να υιοθετεί μια οδηγία που να αντιμετωπίσει το θέμα της ενδοκοινωνικής βίας. Της βίας με βάση το φύλλο, συγγνώμη. Πρόεδρος, ευχαριστώ. μια... Είναι πολύ σημαντικό να διαθέτουμε μια οριζόντια οδηγία και ελπίζω ότι η Δανική Προεδρία, η Δανέζικη Προεδρία θα το αναλάβει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την τόσο ωραία παρουσίαση και την ενδιαφέρουσα έκθεση. Και διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πάντοτε είναι πολύ θετικό να βλέπει κανείς πώς ένα τόσο παλιό και γνωστό θέμα μπορεί κανείς να το χειριστεί με τόσο ενδιαφέρον. Και είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε προχωρήσει καθόλου. Δεν έχουμε κάνει βήματα μπροστά και είναι πολύ ενδιαφέρον και ανησυχητικό να βλέπουμε και πώ ε, και νέε γυναίκε αντιμετωπίζουν το θέμα της ανισότητα τόσο έντονα. Να πω ότι πρόσφατα έγινα και πάλι γιαγιά και πολλά από τα θέματα που ασχολούν ε, την κόρη μου και τις γυναίκες στη ηλικία αυτή είναι πολύ ε, ανησυχητικά η ισότητα δεν έχει επιτευχθεί σε όλους τους τομείς. Καθώς αν έχει κανείς την εκπαίδευση, την ίδια μόρφωση, θα, θα έπρεπε να έχει την, ε, το δικαίωμα στην ίδια απασχόληση και στην ίδια αμοιβή. Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Βλέπουμε λοιπόν πρακτικά τις ανισότητες. Μια γυναίκα επίσης που αναλαμβάνει πολύ μεγάλο μέρος ε, των εργασιών στον οικοκυριό και ταυτόχρονα πολλά άλλα καθήκοντα, βλέπει κανείς πως ακόμη η κοινωνία βλέπει ότι υπάρχουν γυναικείες και ανδρικές δουλειές. Συνεχίζει να υπάρχει αυτή η άποψη και μάλιστα οι δουλειέ στο σπίτι ε, υπάρχουν κοινωνίες που ακόμα τις βλέπουν πολύ αρνητικά ότι σαν αναλαμβάνει ένα άντρα. Συνεχίζουν λοιπόν να υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα. Όταν μιλούμε λοιπόν ε, ίσε αμοιβέ για ίδιε εργασίες πρέπει να ρωτηθούμε τελικά κατά πόσον αναγνωρίζεται ο ρόλος των γυναικών σε όλους τους τομείς. Επίσης, ε, η γυναίκα που μένει στο σπίτι για να φροντίσει τα παιδιά και τους ηλικιωμένους και ποτέ δεν αναγνωρίζεται αυτό το έργο ως εργασία εξίσου σημαντική και με το, ε, αν θέλετε, στο ίδιο επίπεδο όπως μια θέση ενός τραπεζικού. Ε, είναι και αυτό ένα σημαντικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο λοιπόν οι ίσες αμοιβέ και οι ίσες πρόσβαση στην απασχόληση. Έχω την αίσθηση ότι και εμείς οι ίδιες οι γυναίκες δεν το συνειδητοποιούμε πολλές φορές αυτό και όταν συνειδητοποιούμε ένα κάπως αργά στο βίο μας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πολύ περισσότερο τον ρόλο των γυναικών σε όλους τους τομείς και δεν περιοριζόμαστε αποκλειστικά στην απασχόληση και στις αμοιβές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπει κανείς ε, βήματα προόδου σε αυτό το θέμα και ιδιαίτερα η μείωση του χάσματος της ε, αμοιβέ είναι πολύ σημαντικό. Θυμάστε την εξτρατή του 2007, όπου τότε το χάσμα ήταν τη τάξη του 15%. Δηλαδή, οι γυναίκε πρέπει να εργαστούν 54 μέρε και πάνω ενώ τώρα 63 ε, μέρες παραπάνω αν θέλετε βεβαίως ε, έχουν και την ημέρα του στο Μάρτι έτσι, που τις γιορτάζουμε αλλά δεν πιστεύω ότι τελικά αυτό σε τίποτα κατά την Ουγγρική Προεδρία ο Πρωθυπουργό προσυπέγραψε ένα νέο σύμφωνο για τις ε, ίσες ευκαιρίες και τις αμοιβέ, αλλά να πω ότι αυτή η αρχή υπήρχε στην συνθήκη της Ρώμης του 1957 Η Ισπανική Προεδρία ήταν πολύ φιλόδοξη ότι το χάσμα αυτό ε, θα εξαλειφθεί πολύ σύντομα. Τελικά φαίνεται ότι αυτό είναι ρεαλιστικό. Ρεαλιστικό θα ήταν να πούμε να μειώσουμε το χάσμα κατά 1% ετησίως Δυστυχώ. Δεν είναι ήμουν παρούσα στη συζήτηση για τις μεταρρυθμίσεις ε, στο συνταξιτικό σύστημα. Αλλά φοβούμαι ότι όταν υπάρχει χάσμα στις αμοιβές, θα υπάρχει χάσμα και στις συντάξεις. Το έγγραφό σας είναι πολύ σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως ο Επίτροπος Άντορ ναι, προσωπικά καταβάλει προσπάθειες, αλλά τελικά αυτό το θέμα λείπει στην ατζέντα του. Πρέπει αυτόν το κατεστήσουμε κατανοητό. Μιλούμε και για την έννοια των γυναικών. αν δεν εντάξουμε και τη διάσταση του φύλου ε, στο νέο πακέτο για τη μεταρρύθμιση των εξωτερικών συστημάτων, τότε το πρόβλημα της ένδυσης των γυναικών θα οξυνθεί περαιτέρω. Οι γυναίκες άνω των 65 ε, έχουν υψηλότερο κίνδυνο να περιελθούν σε ένδυα. Θα πρέπει λοιπόν να ανεβάσουμε το επίπεδο των κατώτατων συντάξεων και βεβαίως παραγνωρίζουμε συνεχώ και ξεχνάμε συνεχώ το γεγονό τη μη αμοιβόμενη εργασία των γυναικών. Και όπω ε, ορθά είπαν και οι συνάδελφοι, οι γυναίκε εργάζονται συνεχώ στο σπίτι και δεν πληρώνονται ποτέ. Αν πάρει κανεί μια κουβερνάτα στο σπίτι, κοστίζει πολύ περισσότερο, ενώ ε, η γυναίκα είναι δωρεάν. Είναι πολύ σημαντικό να τα αναφέρουμε και όλα αυτά πιστεύω στο κείμενό σας. Το... Η νέα πρόταση για τη μεταρρύθμιση των εξωτερικών συστημάτων είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία τώρα. Η ίση εκπροσώπηση στην διαδικασία πληροφοριών. Είναι πολύ σημαντικό θέμα. Με χαρά άκουσα τον Ορβηγό Πρωθυπουργό πριν από λίγες μέρες να μιλάει για αυτό το θέμα. Και με έπεισε. Αν θέλετε κράτη δικαίου, και πρόνοιας θα πρέπει να βάλετε στο κέντρο της διαδικασία λήψη αποφάσεων τις γυναίκες. Στην Νορβηγία, στον επιχειρηματικό κόσμο της Νορβηγίας, το 40% των ε, θέσεων ε, ευθύνης το έχουν οι γυναίκες. Ναι, το 60% το κρατούν ε, οι άνδρες, αλλά Τελικά αυτό που μας οδηγεί σε μια κοινωνία σε κρίση, αλλά τελικά οι γυναίκες καλούνται σε ένα μεγάλο βαθμό να φέρουν το βάρος αυτής της κρίσης. Είναι όλα στοιχεία που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη επίσης. Όσον αφορά το θέμα της βίας, και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας απασχολήσει περισσότερο. Πιστεύω ότι κάνατε εξαιρετική δουλειά και επίσης ε, η αναφορά στους ε, ομοφυλόφιλου κτλ. είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί ε, είναι κάτι που πρέπει να σεβόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήρθα κάπως αργά ίσως να αναφέρθηκε το θέμα αυτό. Απλώς θέλω να επισημάνω είναι ε, πολύ σημαντικό να έχουμε την ίδια αμοιβή για την ίδια απασχόληση. Πολλές φορές οι γυναίκες έχουν πολύ καλύτερα ε, προσόντα, πολύ περισσότερα προσόντα και πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε τούτο ακριβώς να γίνεται σεβαστό. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Νομίζω ότι η κυρία Βανκέρα από την Κομισιόν θέλει να λάβει το λόγο. Παρακαλώ. Um, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την εισηγήτρια για το πολύ ενδιαφέρον σχέδιο έκθεσης. Υπάρχουν πρωτότυπα σημεία ε, σημεία μάλλον με πρωτότυπο περιεχόμενο και επισύρει την προσοχή μας σε ορισμένα ενδιαφέροντα θέματα. Η ετήσια έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πολύ σημαντικό κείμενο. Συντάσσουμε την έκθεση αυτή από το 2004 και εντεύθεν μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ζήτησε από την Κομισιόν να συντάσσει την έκθεση αυτή σε αιτήσια βάση συνεργασία με τις χώρες μέλη. Και βεβαίως λαμβάνονται υπόψη οι εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για μας τούτο αντιπροσωπεύει ε, μια πολύ σημαντική πηγή πληροφόρησης, διότι το Κοινοβούλιο κάθε χρόνο με τη δική του συμβολή αποτελεί πηγή έμπνευσης για μας, για τη σύνταξη των εκθέσεων αλλά και την εκπόνηση πολιτικών. Θα έχετε παρατηρήσει ότι η έκθεση του 2011 που είναι και το θέμα του σχεδίου έκθεσής σας, ακολουθεί τη νέα δομή. Την στρατηγική ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών 2010-2015 υπάρχει και ένα παράρτημα με στατιστικά στοιχεία. Με πολύ σημαντικά στατιστικά στοιχεία αναφύλλω στατιστικά στοιχεία στα οποία αναφερθήκατε επανειλημμένως σήμερα. 60% των τελειοφύτων των πανεπιστημίων στην Ευρώπη είναι γυναίκες ας πούμε και αυτός ο πίνακα στατιστικών στοιχείων είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Την έκθεση του 2011 διακόπτη, κυρία. Συγγνώμη. Ανέφερα ότι πρέπει να πάω σε μία συνεδρίαση με τον Μάριο Ντράγκη και επειδή θα παρέμβω και εκεί ζητώ συγγνώμη διότι είναι πολύ βάρβαρο αυτό που κάνω αλλά δεν μπορώ να παρίσταμε σε δύο συνεδριάσεις. Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο λοιπόν, λοιπόν και να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι διμερώς θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Απλώς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλα τα σχόλια που έκαναν. Ξέρω ότι υπάρχει περιορισμένο πεδίο κατά το πρώτο σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει οι παρεμβάσεις ήταν πολύτιμες και θα ληφθούν υπόψη υπό μορφή τροπολογιών. Ζητώ πραγματικά συγγνώμη για την παρέμβασή μου αυτή. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, κανένα πρόβλημα, καταλαβαίνω και έπρεπε και εγώ να είχα παρέμβει. Κύριε Μακένη, τώρα έχετε το λόγο, παρακαλώ. Συνεχίστε. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η έκθεση 2011 έχει και ένα άλλο παράρτημα το ε, έγγραφο εργασίας για, τις, ε, για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων από γυναίκες, η συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια εταιριών και αυτό το θέμα ήδη συζητήθηκε στην ε, συζήτηση που προηγήθηκε και το θέμα της συμμετοχής των γυναικών στην λήψη οικονομικών αποφάσεων θα υπάρξει αναφορά το Μάρτιο του 2012 για την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς το θέμα αυτό, δηλαδή η συμμετοχή των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Χαιρετίζουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης που συνέταξε η συγγήτρια, η οποία έφερε επιτάπητος σειρά ενδιαφέρον, ενδιαφερόντων σημείων, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή της οικονομικής κρίσης, διότι γνωρίζουμε ότι η οικονομική κρίση συνεχίζει να επηρεάζει ε, το θέμα της ισότητας ανδρών γυναικών, την αγορά εργασίας κλπ. Η Κομισιόν θα απαντήσει σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία θέτει η έκθεση. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στους στόχους της τις ε, κρεμούσες οδηγίες αλλά και τις νομοθετικές προτάσεις. Επίσης ε, το θέμα των μονογονεϊκών οικογενειών. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσουμε σε αυτά τα επιμέρους ειδικά θέματα. Εν πάση περιπτώσει όμως γενικά για μία ακόμα φορά χαιρετίζουμε την έκθεση αυτή και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Στη φάση αυτή μπορούμε να ολοκληρώσουμε και θα ήθελα να τονίσω το... Να τονίσω ότι έχουμε το εξή χρονοδιάγραμμα. 10 ε, Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα ε, συζητήσουμε τις τροπολογίες στις 25-26 για τις ψηφίσουμε στις 27 Φεβρουαρίου και θα έρθει στην Ολομέλεια του Απριλίου. Και τώρα περνούμε στο σημείο 6 της σημερισίας διατάξεως. Ε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα πάρα πολύ καλά γιατί σκεφτόμουν κάτι άλλο. Ποια είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες? 10 Ιανουαρίου? Ναι, 10 Ιανουαρίου. Λοιπόν, σημείο 6. Ενεργειακή απόδοση και κατάργηση των οδηγιών κλπ. κλπ. Θα δώσω το λόγο στην Τρέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την απουσία μου στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης. Ήμουν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που λαμβάνει χώρα ταυτόχρονα και χρειάστηκε να παραστώ εκεί γιατί ήταν εκεί παρούσα η Επιτροπή κυρία Δαμανάκη. Πρέπει λοιπόν ε, να είμαστε πανταχού παρόντε, ε, να τρέχουμε από τη μία επιτροπή στην άλλη. Πάντως σας πω ότι αύριο ε, θα συμβεί το ίδιο πάλι. Και μάλιστα είμαι σκιώδη ηγητή. για το θέμα των γυναικών και της κλιματικής αλλαγής που μετακινήθηκε για αύριο. Και αυτό είναι πρόβλημα για μένα διότι αύριο πρέπει να ψηφίσω στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Είναι δύσκολο να συμμετέχουμε σε δύο επιτροπές ταυτόχρονα. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ενεργειακής απόδοσης και κατάργηση των οδηγιών 2004-8 και 2006-32. Δύο λόγια για ε, το πλαίσιο αυτής της οδηγίας. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, καθόρισε ε, το στόχο του 10% ε, εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2020 και αυτό αποτελεί ένα από τους πέντε βασικούς στόχους της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την ευφυή e e, βιώσιμη και συμπεριληπτική ανάπτυξη. Σύμφωνα με τις αξιολογήσεις εκτιμήσεις κομισιών που λαμβάνουν υπόψη ε, τις εθνικούς στόχους και τις εθνικές πολιτικές που έχουν καθορίσει τα κράτη-μέλη στο πλαίσιο της στρατηγικής Ευρώπη 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φτάσει στο 50% του στόχου του 20% μέχρι το 2020. Αυτή η πρόταση οδηγίας καθορίζει ένα κοινό πλαίσιο για την πρόθεση της ενεργειακής αποδοτικότητας ε, Τη ενεργικής απόδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε τελικά να, είναι, να καταστεί δυνατή επίτευξη του στόχου της εξοικονόμηση κατά 20% μέχρι το 2020 έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια αυξημένη ενεργειακή απόδοση ε, και για την περίοδο μετά το 2020. Καθορίζει κανόνες για την απάλληψη των εμποδίων και την διόρθωση ορισμένων αδυναμιών της αγοράς που παρεμποδίζουν την απόδοση στην προμήθεια και τη χρήση της ενέργειας. Ορισμένες διατάξεις περί ε, των οδηγιών 2004 ε, και 2006 θα καταργηθούν. Αυτή η πρόταση οδηγία ε, μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία προκειμένου να υπογραμμίσουμε μια ακόμα φορά την σημασία της πρόσβασης των γυναικών σε εξειδικευμένη κατάρτιση προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους ε, της ενεργειακής απόδοσης και προκειμένου να δώσουμε στις γυναίκες τη δυνατότητα να καταλάβουν μελλοντικέ θέσει εργασία στου τομεί του ε, συναφεί με την ενεργειακή απόδοση. Μια άλλη πτυχή που υπογραμμίζω σε αυτή την έκθεση είναι ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προωθήσουν έναν κοινωνικό στόχο στα μέτρα τα οποία θα λαμβάνουν για την ε, επιτυχία του ενεργειακού στόχου μέσω της συμπερίληψης μέτρων που θα εφαρμόζονται στην, ε, στα νοικοκυριά τα οποία πλήττονται από την ενεργειακή ένδια. Θα χρειαστούν κίνητρα και μέτρα για, κοινωνικές, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες έτσι ώστε αυτές οι ομάδες να ε, βελτιώσουν την ενεργική απόδοση στα σπίτια τους και ταυτόχρονα να, μειωθούν, ε, να μειωθεί το κόστος της ενέργειας. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να σχεδιαστούν λαμβάνοντας υπόψη το φύλλο, τη διάσταση φύλλου και εκεί βέβαια μπαίνει η δική μας αρμοδιότητα. 13 προτάσεις τροπολογίας κατατέθηκαν. Κατά την άποψή μου η πλειοψηφία τους είναι θετικές, εμπλουτίζουν τη θέση της Επιτροπής μας με την εξαίρεση το, της 14 και 21 ε, που υπερβαίνουν το τομέα αρμοδιοτήτων μας. Γι' αυτό το λόγο και θα τις καταψηφίσω. Επαναλαμβάνω τις τροπολογίες 14 και 21 που δεν μπορούν να ενταχθούν στο πεδίο της δική μας Επιτροπής. είναι θεμητέ, είναι λογικέ, αλλά μάλλον αντιστοιχούν περισσότερο στι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Βιομηχανία ή τη Επιτροπή Περιβάλλοντο, όχι στι αρμοδιότητε τη Επιτροπή Γυναικών. Σε ό,τι αφορά τι άλλες προτάσει, όμω μπορώ να ε, συμφωνήσω με θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγητρία. Κυρία Κλάς, παρακαλώ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την ε, συνάδελφο, την Εστρέλα, για την γνωμοδότηση και την όλη παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το ευρύτερο πλαίσιο πλέον μιλούμε για ενεργειακή απόδοση. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει αυτή η συνειδητοποίηση από όλου μα. Η συνάδελφο, η κυρία Στρέλο, έθεσε αν θέλετε, στο επίκεντρο τους ε, κλιματικού ε, στόχου εν ώψη του 2020. Θα ε, έλεγα όμω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια άλλη διάσταση, διότι διαφορετικά καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο σημείο. Θέλουν μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση στην κατανάλωση ενέργεια. Όμω, λέω ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα πρέπει να έχει και ως στόχο την αντιμετώπιση της ένδυας, ε, της ε, ε, πείνας και καλύτερη χρήση των πόρων του πλανήτη. Ειδικά η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη εν γέννη αντιμετωπίζουν βαρετική ένδυα ενδιακούς πόρους. Λαμβάνοντα υπόψη την αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού, πρέπει να κάνουμε κάτι, διότι θέλουμε η ανάπτυξη να συμπεριλαμβάνει όλο το παγκόσμιο πληθυσμό, ώστε να υπάρξει ευημερία και υγεία για τον πληθυσμό του πλανήτη. Αυτά είναι κρίσιμη σημασία θέματα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε καλύτερη διαχείριση των πόρων και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε περισσότερες διακασίες σε αυτό το τομέα. Η Επιτροπή στην ομοθέτησή της ζητά περισσότερη πληροφόρηση, ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις ορθές υπερηφορές, την σωστή κατανάλωση κτλ. Συνεργασία των κρατών μελών προκειμένου. Θυμάμαι πάμπολες συζητήσει και στο παρελθόν ε, για το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη συνηθίζουν να είναι πολύ επιφυλακτικά σε αυτό το τομέα. Όμως, έχουμε και το δικαίωμα να υπενθυμίζουμε συνεχώς ότι τα κράτη-μέλη έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση να κάνουν κάτι η ενημέρωση σήμερα είναι πάρα πολύ εύκολη. Ξεκινά από το σχολείο, καταλήγει στο διαδίκτυο και υπάρχει παντού. Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε σε μια καλύτερη ενεργειακή απόδοση. Και εδώ η διάσταση της γυναίκας είναι πολύ σημαντική, διότι η γυναίκα στο σπίτι, στο νοικοκυριό είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Η γυναίκα είναι συνήθως αυτή που αποφασίσει και τον καλύτερο τρόπο θέρμανσης ε, υψήξης του σπιτιού. Παρά τα αυτά βλέπουμε ότι αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη. Το 18% της ε, κατανάλωσης ενέργειας γίνεται στα νοικοκυριά. Και πραγματικά όταν έχουμε σπίτια με κακή μόνωση είναι κατασπατάληση ενέργειας. Χάνεται η ενέργεια. Και δύο είναι οι σημαντικοί πυλώνες. Καλύτερη μόνωση και ε, η σωστή κατασκευή νεόπιτων κατοικιών. Έπειτα, η εκπαίδευση, η αγωγή των παιδιών και αυτό εξαρτάται από τη γυναίκα. Η γυναίκα με την σωστή ευφυή χρήση της ενέργειας διδάσκουν τα παιδιά το ίδιο και στους παιδικούς σταθμούς και στα σχολεία. Εκεί μαθαίνουν τα παιδιά. Εκεί θα αρχίσουν να ενημερώνονται οι μελλοντικοί χρήστες για την κατανάλωση που θα κάνουν αύριο. Άρα λοιπόν η γυναίκα έχει ένα ρόλο κλειδί προκειμένου και ένα ρόλο που ξεπερνά τα όρια του νοικοκυριού. Ξέρουμε ότι η γυναίκα εργάζεται και συμμετέχει και στη διαδικασία των αποφάσεων για την καλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Και αποφασίζουν και σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, περιφερειακής αυτοδιοίκησης. Η ενεργειακή απόδοση είναι κάτι που απασχολεί σε όλα τα επίπεδα ε, διακυβέρνησης και άρα οι γυναίκες πρέπει να έχουν πρώτο λόγο εν προκειμένου. Στηρίζω ε, το σχέδιο γνωμοδότησης ε, της κυρίας Εστέλα και την ε, προσέγγιση που έκανε επί του θέματος. Από ό,τι βλέπω τώρα, όσον αφορά τις τροπολογίες, έχει και η συγγήτρια κάποια ερωτηματικά. Συμμερίζομαι και εγώ αυτά τα ερωτηματικά για κάποιες ε, τροπολογίες, διότι Κάποια θέματα δεν υπάρχουν αρμοδιότητε. Υπάρχουν βεβαίω και άλλε τροπολογίε που πρέπει να γίνουν, διότι βλέπουμε ότι το κείμενο τη Κομισιόν είναι πάρα πολύ διστακτικό, καλή και ενθαρρύνει η Κομισιόν τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι, γενική απόδοση. Εμεί θεωρούμε ότι θα πρέπει ε, να είναι πολύ πιο δεσμευτική η διατύπωση. Ε, θέλω να αναφερθώ στην τροπολογία 11, την οποία θεωρώ σημαντική. Όσον αφορά τις περιφέρειες, ε, και την ε, περιφερειακή προσέγγιση. Δεν την καταλαβαίνω απόλυτα αυτή την τροπολογία θα έλεγα. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο μέτρο μα αναλογή. Θέλουμε απόδοση και αποδοτικότητα σε όλα τα επίπεδα. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώ το νόημα αυτής της τροπολογίας. Πιστεύω ότι όλοι πρέπει να κάνουν το μερίδιο που του αναλογεί στο μέγιστο βαθμό που μπορούν. Πιστεύω ότι αύριο πρέπει να υπερψηφίσουμε το σχέδιο γνωμοδότηση, ίσω με κάποιε μικροαλλαγέ. Αύριο θα είμαστε εδώ παρόντε στη ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Τόμσον. Ε, Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ και εγώ την εισηγήτρια για αυτή τη γνωμοδότηση. Είναι πολύ ε, σημαντικός ο τομέας και ε, θίγεται πολύ σημαντικές πτυχές του. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί σήμερα ξεκινήσαμε συνεδρίαση με την παρέμβαση του Επιτρόπου Άντορ, ο οποίος μας είπε ότι στα κράτη-μέρη υπάρχει έλλειψη κατανόησης του θέματος της ε, συνεκτίμησης διάστασης του φύλου στις πολιτικές. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε στο τραπέζι αυτή την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση αλλά δεν βλέπουμε πουθενά τη διάσταση του φύλου εδώ. Άρα δεν υπάρχει το πρόβλημα μόνο σε επίπεδο μελών. Θα έλεγα μάλιστα ότι ο Επίτροπο στην αρχή μα είχε υποσχεθεί να αναλάβει μια πρωτοβουλία για να καταρτιστεί ένας χάρτης για την ενσωμάτωση του, της διάστασης του φύλου στις πολιτικές και αυτό έγινε στις 11 Μαρτίου 2010. Προσυπέγραψαν αυτή την πρωτοβουλία όλοι οι επίτροποι, ώστε σε όλες τις προτάσεις τους να συμπεριλαμβάνουν τη διάσταση του φύλου. Εδώ ε, δυσκολεύομαι να δω πώς εντάχθηκε η διάσταση του φύλου σε αυτή την πρόταση. Ουσιαστικά οι γυναίκες είναι πλέον υπεύθυνε για τον τρόπο ενεργικής κατανάλωσης ε, στα νοικοκυριά. Επίσης είναι οι γυναίκες αυτές που κατά κύριο λόγο διαχειρίζονται τα οικονομικά του νοικοκυριού. Να λοιπόν ένα καλό παράδειγμα μιας πρότασης όπου θα μπορούσε να μας δείξει τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα της διάστασης του φύλου. Επίσης στην οδηγία αυτή μιλούμε πολύ συχνά για την ενεργειακή ένδυα. Ποιοι εκπροσωπούν την ενεργειακή ένδυα στην Ευρώπη, οι γυναίκες, η ένδυα στην Ευρώπη έχει ένα πρόσωπο και αυτό είναι γυναικείο. Στο Ενωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, πολλά νοικοκυριά που αποτελούνται από ένα μόνο δεν έχουν απλά πρόσβαση στην ενέργεια γιατί είναι πάρα πολύ ακριβή. Η μόνωση λοιπόν των σπιτιών που είναι το τόσο σημαντικό, θα έλεγα ότι πλέον ενδεεί στην κοινωνία μας είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν σήμερα το πρόβλημα και άρα με την νέα πρόταση θα πρέπει να αποφεληθούν και οι γυναίκε είναι μεταξύ αυτών. Θα πρέπει λοιπόν και στην ηλικιακή απόδοση να ε, συμπεριληφθεί υπόψη η διάσταση ε, του φύλου. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή την γνωμοδότηση που εκπονεί η Επιτροπή μας. Τώρα, κάτι άλλο όσον αφορά τις εργασίες στον ενεργειακό τομέα. Βλέπουμε ότι οι περισσότερες θέσεις εργασίας καλύπτονται από άντρες στον τομέα. Και αυτό τι μου θυμίζει. Όταν ο Κέν Λίβνιστον ήταν δήμαρχος στο Λονδίνο, απέδειξε ότι οι πιο πολλοί χρήστες του μετρό ήταν γυναίκες. Αντιστρόφω όμως ανάλογα τον ποσοστό των εργαζομένων γυναικών στο μετρό. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να διασφαλίσουμε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και για τις γυναίκες και πιστεύω ότι ε, μια καλή ευκαιρία είναι για αυτή η πρόταση οδηγίας. κυρία Γκραμαή έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι που λαμβάνω το λόγο μετά την κυρία Τόμσον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στράλη για την γνωμοδότηση. Η συνάδελφος ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό. Τούτο ήταν μέρος της ε, εκστρατείας, της εκλογικής εκστρατείας του 2009. Το Μάρτιο του 2010 εγκρίθηκε ένα έγγραφο από την Επίτροπο Βιβιαν Ρέντινγκ. Το έγγραφο αυτό με μεγάλη σαφήνεια ανέφερε ότι κάθε Επίτροπος πρέπει να λαμβάνει υπόψη το θέμα της ισότητας των δύο φύλων και την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας στις δραστηριότητές του και διαπιστώνουμε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά και δίνουμε ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, σε αυτή την Επιτροπή. Με τη γνωμοδότηση η συγγήτρια είχε τη δυνατότητα να επισημάνει το ρόλο των γυναικών και το, ιδιαίτερα στο θέμα της κατάρτισης για να επιτευχθεί ο, ο στόχος της ενεργειακής απόδοσης. Νομίζω ότι μιλούμε για ένα ιστορικό δικαίωμα ε, στο παρελθόν θέλαμε τα σπίτια να είναι πολύ ζεστά. Στις μέρες μας όμως όταν ε, η θερμοκρασία φτάνει 24-25 βαθμούς ε, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε χαμηλότερα επίπεδα. Όταν πρώτο φτάσαμε στις Βρυξέλλες το 2004 ένας από τους συναδέλφους έλαβε μια επιστολή Μία από τις συναδέλφους έλαβε επιστολή η οποία ανέφερε ότι έκανε υπερβολική κατανάλωση ενέργειας και θα έπρεπε να τη μειώσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συμβεί παντού και σε κάθε χώρα μέλος. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία εμείς μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε για να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Και νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε από πολύ νωρίς από τον υπηαγωγείο. Τα παιδιά πρέπει να κατανοήσουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση είναι κάτι πολύ σημαντικό. Η Ρίτα Τόμσον πολύ ορθά επεσήμανε ότι η φτώχεια και η ενεργειακή ένδια συνδέονται με, με το θέμα των γυναικών και πιστεύω και ελπίζω ότι η Επιτροπή αυτή θα λάβει υπόψη την άποψη αυτή πολύ σοβαρά και ελπίζω ότι θα δεχθούμε, θα εγκρίνουμε αυτή τη θετική προσέγγιση. Ο Πρόεδρος. Και θα ήθελα τώρα να λάβω το λόγο εγώ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόταση, ε, πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπάρχει η διάσταση της ισότητας, να ενσωματώνεται η διάσταση της ισότητας των φύλων στα πάντα. Και δεν είναι η μόνη πρόταση, έχουμε δύο τέτοιες προτάσεις. Δεν θα μακρηγορίζω. Υπάρχουν δύο προτάσεις για, για τις 15 και 18. Διότι η προσέγγιση είναι ορθή, αλλά ο τρόπος διατύπωσης ή σύνταξη, το εμφανίζει ε, σαν να υπάρχει κάποιος ε, βιολογικός λόγος. Άρα λοιπόν η τροπολογία 18 είναι ένα χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα διότι μιλά για την αρμοδιότητες των γυναικών στον οικοκύριο. Συμφωνώ ότι σε πολλές περιπτώσεις οι γυναίκες έχουν την ευθύνη για την λειτουργία του νοικοκυριού και συνεπώς <laughs> έχουν αρμοδιότητα από αυτού αλλά αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι είναι γυναίκες οφείλεται στη κοινωνική τους θέση δεν θέλουμε να ηχεί ως μια αρμοδιότητα που προκύπτει από τη βιολογική διάσταση ας πούμε της γυναίκας ένα δεύτερο σημείο που δύσκολα θα ψηφίσω ε, υπέρ λοιπόν είναι ακριβώς αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος. Ο κύριο Άψον έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι συμφωνώ με την κυρία Κλάς. Να πω καταρχήν ότι κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι αυτά είναι δευτερεύοντα και τετριμένα, ότι έχουν να κάνουν με τίποτα λαμπάκια και διακόπτες κλπ. Αλλά αν δεν αντιμετωπίσουμε αυτά τα πράγματα σωστά φοβούμε ότι θα αποτύχουμε παντού. Από εδώ πρέπει να ξεκινήσουμε. Ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει επαρκή και σωστή πληροφόρηση σχετικά με, την, ε, με τα ενεργειακά όπως επίσης και τις αποδόσεις και επιδόσεις των συσκευών που χρησιμοποιεί. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι γυναίκες εμπλέκονται πολύ περισσότερο. Είναι ε, τομέας πολιτικής που συνδέεται άμεσα με τα νοικοκυριά, με τα σπίτια και ιδιαίτερα σε περιόδους ε, αυξημένων τιμών της ενέργειας. Όταν ε, μιλούμε για ενεργειακή πολιτική ε, αναφερόμαστε πολύ συγκεκριμένα και κατά κύριο λόγο στη θέρμανση, όπως είπε και η κυρία Κράσα. Είναι λοιπόν ένας πολύ σοβαρός τομέας και χαίρομαι που επισημαίνεται ότι πρέπει να επιτύχουμε αυτό το στόχο του 20%. Και όπως επισημαίνει η κυρία Τόμψον, σίγουρα υπάρχει πεδίο για δημιουργία πολλών θέσεων απασχόλησης. Ε, κατά το παρελθόν πρόκειτο για δουλειές, για απασχόληση κατά κύριο λόγο ανδρική. Ενώ αυτή τη στιγμή Μιλούμε για κάτι άλλο, μιλούμε για βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομένων και σίγουρα αυτό θα λάβει υπόψη και την ε, διάσταση της ισότητας. Δεν θέλω να κάνω άλλα σχόλια παρά μόνο να ε, επισημάνω θετικά τα όσα λέγονται. Αναφέρομαι ειδικά στην τροπολογία 17 που περιορίζει το επίπεδο της φιλοδοξίας μας ας πούμε από 1,5% σε 1% ε, έχω δυσκολία λοιπόν να υιοθετήσω την πρόταση αυτή η οποία έρχεται σε αντίθεση με τις προσπάθειες που καταβάλουμε. Πάντως ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι αύριο θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Ευχαριστώ λέει η κυρία Στρέλα. Ε, ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για όλα αυτά τα σχόλια, τις παρατηρήσεις. συμμερίζομαι τις ανησυχίες κυρίας Κλάς. Πολύ δε περισσότερο που είμαι μέλος Επιτροπής Περιβάλλοντος, εδώ και δύο θητείες. Συνεπώς ε, είμαι πολύ εξοικειωμένη με έννοιες όπως η ενεργειακή απόδοση. Πέραν αυτού, εγώ υποστηρίζω μια κοινή ενεργειακή πολιτική. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πολλά να κερδίσει αν διαθέτει κοινή ενεργειακή πολιτική. Όχι μόνο διότι θα το περισσότερη ασφάλεια εφοδιασμού και μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην, σε ό,τι αφορά τις πηγές από τις οποίες προμηθευόμαστε ενέργεια, αλλά και γιατί πιστεύω ότι θα εξασφάλιζε μεγαλύτερες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, βέβαια, στην γνωμοδότησή μας δεν τίθεται αυτό ε, το θέμα. Μας ε, ξεπερνάει η κοινή ενεργειακή πολιτική, ξεπερνάει το πεδίο αυτή της έκθεσης της Επιτροπής μας. Εμείς αυτό που ζητούμε είναι να ενταχθεί και η πτυχή του φύλου στον τομέα της ενεργειακή απόδοσης. Συμφωνώ με τα όσα ελέγχθησαν σε ό,τι αφορά την αλλαγή στις ε, συμπεριφορές, στην καθημερινή συμπεριφορά, που ε, αλλαγές που θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε σημαντική αύξηση της ενεργικής απόδοσης. Όλοι μας μπορούμε να συνεισφέρουμε για την επιτυχία του στόχου της ενεργειακής απόδοσης, ε, σβήνοντας τα φώτα όταν δεν είμαστε στο δωμάτιο, όταν δεν χρειάζονται, χρήση ειδικών λαμπτήρων με μεγάλη διάρκεια ζωής και μικρή, μικρότερη κατανάλωση. Ε, αποφυγή ε, συνεχούς χρήσης της θέρμανσης και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να δώσουμε παράδειγμα για τέτοιου είδους συμπεριφορές. Μερικές φορές βέβαια δίνουμε το κακό παράδειγμα. Για παράδειγμα ε, θερμαίνουμε υπερβολικά τις αίθουσες κατά την άποψή μου και σπαταλάμε ενέργεια. Τώρα, σχετικά με τις ε, τροπολογίες τις οποίες αναφερθήκαμε. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην 15 και την 18. Εγώ τις υποστηρίζω όχι γιατί υπάρχουν ε, όχι γιατί η γυναίκα έχει αυτές τις ευθύνες για βιολογικούς λόγους, όχι. Ε, δεν υπάρχουν τέτοιοι βιολογικοί λόγοι. Απλά η κοινωνία αποδίδει μεγαλύτερες ευθύνες στην γυναίκα σε ό,τι αφορά τη, τις, τα οικιακά της καθήκοντα. Το ίδιο με τη μόρφωση των παιδιών, με την φροντίδα των ηλικιωμένων, των ασθενών κλπ. Πρέπει να αλλάξουμε τις συνειδήσεις έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε μια πραγματική ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και σε αυτά τα καθήκοντα. Το σημείο αφετηρίας όμως είναι η πραγματικότητα και αυτήν θα πρέπει να αλλάξουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τροπολογία 17, στην οποία αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, ε, έχει αποσυρθεί. Ακριβώς διότι Ε, ήταν λιγότερο φιλόδοξη από την πρόταση της Κομισιόν. Προφανώς αυτό δεν θα ήταν πολύ ευχάριστο από πλευράς του Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες και υποτίθεται πρέπει να πηγαίνει πιο μακριά. Ακόμα και αν δεν θέλουμε να πάμε πιο μακριά δεν είναι δυνατόν να είμαστε πιο, μάλλον λιγότερο φιλόδοξοι από η ίδια η Κομισιόν. Γι' αυτό η προτείνουσα την απέσυρε τελειώνω λέγοντας ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ζήτημα της πληροφόρησης και της κατάρτισης. Γιατί χωρίς ε, πλήρη πληροφόρηση και κατάρτιση δεν μπορούμε να κάνουμε ελεύθερα τις επιλογές μας. Μόνο έτσι μπορούμε να συμμετάσχουμε ενημερωμένοι και ενημερωμένες στη λήψη των αποφάσεων και μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε τις νέες θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν ε, από την προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας. Ελπίζω ότι και αύριο θα καταφέρουμε με μια ευρία πλειοψηφία να εγκρίνουμε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Στρέλα. Μια διευκρίνηση μόνο να κάνω. Θα ψηφίσουμε αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης αύριο. Ναι. Αυτό που είπατε για την ε, κοινωνική κατασκευή και τη βιολογική κατασκευή, ναι, είναι κάτι που χρήση μια εισβάτηση, γιατί ούτε εσείς γνωρίζετε, ούτε εγώ γνωρίζω απόλυτα όλες τις διαστάσεις και θα πρέπει να δούμε και το θέμα της επιλογής των ειδών. Υπάρχουν κάποια κοινωνικά ε, στερεότυπα που ε, συνεχώς ε, συνεχίζονται και πιστεύω ότι η θεωρία του Δαρβίνου είναι αυτή που θα πρέπει να μας απασχολήσει και να είναι ένα κομμάτι της συζήτησής μας. Ε, να απαντήσω εγώ, λέει ο Πρόεδρος, μήπως αυτό το σχόλιο. Γιατί θα μου πάρει πολύ περισσότερο από ένα λεπτό είναι πολύ γενικότερη συζήτηση που ανοίγεται. Και εγώ δεν ήθελα τώρα να πούμε σε τέτοια συζήτηση. Συνδέεται αυτό το θέμα το πώς βλέπει ο καθένας την πραγματικότητα. Καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε λέξεις που μας παγιδεύουν σε συγκεκριμένα στερεότυπα. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτή τη ζήτηση εδώ, γιατί Ιδάλλως δεν τελειώνουμε ποτέ. Θα ψηφίσουμε, επαναλαμβάνω, αύριο για αυτή την γνωμοδότηση, οπότε αφήνουμε αυτό το σημείο και πάμε στο σημείο 8. Αντιπροσωπή της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών και Ισότητας των Φίλων στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη. 1η ως 4 Νοεμβρίου. Εγώ και η κυρία Άμστερτο Άλντε και κυρία Σινκλέρ από τους διαγεγραμμένους, ε, η κυρία Κιλ Νίλσεν από τους πράσινους, τέσσερις λοιπόν ε, ήμασταν που συμμετείχαμε σε αυτή την αντιπροσωπεία και είχαμε και άλλα δύο μέλη, τον κύριο Μπέλτερ ε, πρόεδρος αντιπροσωπείας για το Ισραήλ και κυρία Μαρκρέτα των Πρασίνων αντιπρόεδρος αντιπροσωπείας για το Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο. Οπότε δεν χρειάζεται να πω το σχετικό έγγραφο που σας ενημερώνει για αυτή την επίσκεψη. Εκεί θα δείτε όλες τις λεπτομέρειες. Ο στόχος ήταν να δούμε το θέμα των γυναικείων δικαιωμάτων και στα Παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ. Την πρώτη μέρα της επίσκεψης είχαμε συνάντηση με προσώπους της Αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη. Επίσης είχαμε συνάντηση με εκπροσώπους ε, γυναικείων οργανώσεων. Τη δεύτερη ημέρα ήμασταν στη Λωρίδα της Γάζας. Συνήθως είναι δύσκολη πρόσβαση στη Λωρίδα της Γάζας, όμως καταφέραμε να πάμε εκεί και να επισκεφτούμε και ένα σχολείο φιλέων. Μπορεί να σας ακούγεται κάτι τετριμένο, αλλά ε, και μόνο το γεγονός ότι υπάρχουν ε, χωριστά σχολεία αρένων και Θηλαίων λέει κάτι. Υπάρχει, μιλάμε για μια περιοχή όπου ε, πολύ συχνά οικογένειες δεν αφήνουν τα κορίτσια να πηγαίνουν σχολείο. Μιλάμε λοιπόν για ένα ιδιαίτερο σχολείο, ένα σχολείο θηλαίων που προσφέρει μόρφωση στα κορίτσια. μόρφωση αλλά και ενημέρωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι πραγματικό παράδειγμα προς μίμηση αυτό το σχολείο. Και ρωτήσαμε και αυτά τα κορίτσια κατά πόσον αυτά τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικαιωμάτων γυναικών είναι κάτι που ζητούν και στο σπίτι και μας είπαν πως ναι, είναι ένα θέμα που έχουν ζητήσει και στο σπίτι. Ε, Έπειτα την ίδια ημέρα είχαμε ε, συνάντηση και με πολλές άλλες οργανώσεις. Τώρα τα περνάω λιγάκι γρήγορα αυτά τα θέματα. Μπορείτε να τα δείτε, όπως είπα, στο έγγραφο. Ε, την επόμενη ημέρα ήμασταν στην Κνέσσετ και είχαμε επαφές με τον πρώτο της Επιτροπής για, το, τη θέση των γυναικών όπως επίσης και με την πρόεδρο της Υποεπιτροπής για την ε, για το εμπόριο γυναικών. Εκεί ακούστηκαν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, βεβαίως και πολύ ανησυχητικά για το θέμα της σωματεμπορίας. Σε επαφές μας με μια άλλη επιτροπή για τα γυναικεία δικαιώματα, συζητήσαμε το θέμα της άδεια μητρότητα. συζητήθηκε το θέμα της γονικής άδεια εν γέννη και της πατρικής δηλαδή άδεια. Θα τρέχω, επαναλαμβάνω πάλι τα θέματα γρήγορα, μετά είχαμε μια επαφή με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Εθνικής Αρχής και να πω ότι μια ενδιαφέρουσα στιγμή ήταν όταν ετέθη το ερώτημα κατά πόσον ε, θα μπορέσουν να ασκήσουν πρακτικά και τα ε, δικαιώματά τους οι γυναίκες, ειδικά σε μια περιοχή ε, σειράξεων. Η απάντηση που λάβουμε από τον Παλαιστίνο Πρωθυπουργό ήταν εν είδη αστεϊσμού ότι αυτή τη στιγμή οι άντρε δεν έχουν καταφέρει τίποτα τόσα χρόνια. Καλό είναι να του βάλουμε στην άκρη και να βάλουμε τι γυναίκε στην εξουσία. Έπειτα είχαμε επαφές με προσώπους της Παλαιστινιακής κυβέρνησης, με πέντε υπουργούς συγκεκριμένα, πέντε γυναίκες υπουργούς. Ε, είχαμε τη χαρά να έχουμε συνάντηση την Υπουργό Γυναικείων Υποθέσεων, Κοινωνικών Υποθέσεων, την Υπουργό Πολιτισμού, την Υπουργό Παιδείας και την Υπουργό Τουρισμού. Και είχαμε μία μακρά συζήτηση για μία πλειάδα ζητημάτων. Από ό,τι θυμάμαι, 25 πέντε υπουργοί αποτελούν το Υπουργικό Συμβούλιο της Παλαιστινιακής Αρχής και πέντε εξ αυτών είναι γυναίκες. Και η βραδιά έκλεισε με ένα δείπνο εργασίας που διοργάνωσε η κυρία Τζάνατ Μαχαήλ που είναι η δήμαρχος της Ραμάλα. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά αυτή η αποστολή ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, ήταν έντονη και γεμάτη ε, επαφές, συνεδριάσεις. Ξεκινούσε ε, νωρίς το πρωί η δουλειά και κατέληγε πολύ αργά το βράδυ. Και αν πρέπει να συνοψίσω αυτή την επίσκεψη σε ελάχιστα λόγια, θα έλεγα ότι το θέμα της ισότητας των φίλων είναι πολύ ζωντανό και ανοιχτό θέμα οπουδήποτε στον κόσμο, και στο Ισραήλ και στα Παλαιστινιακά εδάφη. Η ανάγκη να ενισχυθούν περαιτέρω τα δικαιώματα των γυναικών είναι κάτι που απασχολεί και εκεί. Και θα έλεγε κανείς ότι εκεί οι ανισότητες είναι σε διάφορα στήματα και, και σε διάφορους βαθμούς. Βεβαίως, αυτή τη στιγμή ε, η Παλαιστίνη είναι μια χώρα υποκατοχή, Κατανοείτε πως αυτό επηρεάζει βεβαίως πολύ αρνητικά και τα δικαιώματα των γυναικών. Νομίζω ότι καλό είναι να σταματήσω εδώ, να δώσω το λόγο στην κυρία Νίλσεν που ήταν και μέρος της αντιπροσωπείας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα απλώ να πω, καταρχήν σχετικά με τις γυναίκες ε, στην πλευρά της από πλευράς Παλαιστίνης. Αυτό το οποίο είδαμε είναι αρκετά παράδοξο. Από τη μία πλευρά είναι αληθές ότι οι Παλαιστίνιες όπως και πολλές άλλες στον κόσμο ζουν σε μια πατριαρχική κοινωνία άρα λοιπόν υφίστανται την καταπίεση που οφείλεται στην πατριαρχική κοινωνία αλλά υπάρχει και η δεύτερη καταπίεση που είναι οι συνέπειες της ε, ε, ε, απεικιοκρατίας στην Γάζα, στη Γάζα συγγνώμη, υπάρχει ακριβώς αυτή η πατριαρχική κοινωνία αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ο αποκλεισμός. Αποκλεισμός ο οποίος έχει σοβαρές δραματικές ανθρωπιστικές συνέπειες. Πάνω από το 50% του πληθυσμού που αποτελείται από παιδιά, από ανήλικα, παιδιά, οι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για να αγωνιστούν για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα υποκαθεστώς αποκλεισμού. Άρα λοιπόν η κατάσταση των γυναικών στη Γάζα είναι φοβερή. Το γνωρίζαμε αυτό πριν πάμε βεβαίως. Ενώ στην... Ε, en même temps, euh, ce qui est intéressant avec les Palestiniens, c'est qu'on découvre στη θετική όχθη του Ιορδάνη και εκεί διαπιστώνει κανείς ε, ότι υπάρχει ένα σημαντικός αριθμός γυναικών με υψηλή μόρφωση. Και πράγματι συναντήσαμε πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν ε, εκπαίδευση και κατάρτιση υψηλή. Άλλο παράδοξο. Η ανεργία. Είναι γεγονός τόσο για, για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες εδώ λοιπόν παράδοξα τα οποία αντιμετωπίζει κανείς. Από την άλλη υπάρχουν οι κρατούμενοι. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Χθε μόλις είδαμε ένα δεύτερο κύμα απελευθέρωσης κρατουμε... Παλαιστινίων κρατουμένων. Αυτή τη φορά δεν ε, συναντήσαμε ενώσεις οργανώσεις ε, γυναικών. Με άλλη ευκαιρία είχαμε τη δυνατότητα αυτή. Οι Παλαιστίνιες λοιπόν έχουν πολλές δυσκολίες στο να επισκέπτονται τους ε, κρατούμενους ε, άνδρες γιους διότι πάρα πολλά νεαρά παιδιά, αγόρια ε, βρίσκονται στις φυλακές και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες, ταπεινώσεις, δυσκολίες. Αυτό όλα αποτελούν την καθημερινότητα των Παλαιστινίων γυναικών που έχουν κρατουμένους άνδρες ή παιδιά. Από την πλευρά τώρα των Ισραηλινών. Υπάρχουν γυναίκες οι οποίες πραγματικά εμπνέουν ελπίδα. Συναντήσαμε εκπροσώπους της Ένωσης Watch που είναι Ισραηλινές, Ισραηλινές που μάχονται, που αγωνίζονται ακριβώς για την, για την ε, ε, κατάργηση των παραβιάσεων και της βίας που ασκείται εναντίον των ε, Παλαιστινίων, κυρίως στα checkpoints. Είναι οργανώσεις γυναικών ή κατά κύριο λόγο γυναικών που αγωνίζονται ακριβώς υπέρ των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων. Οι γυναίκες ξέρετε ότι υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία στο Ισραήλ και όλο και περισσότερες εγγράφονται σε, έναν, μια οργάνωση που αποκαλείται μαχητές για την ειρήνη. Από πλευράς δηλαδή Ισραηλινής υπάρχει ακριβώς αυτή η ελπίδα που βγαίνει μέσα από τις οργανώσεις των γυναικών. Αυτό ήθελα να προσθέσω στα όσα είπε ο Πρόεδρος. Είναι ένα σημείο το οποίο πράγματι θα υπάρξει και στην έκθεση. Στο Ισραήλ ακούσαμε πολύ να ομιλούν για το θέμα του γάμου. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται πολιτικός γάμος στο Ισραήλ και υπάρχουν πολλά προβλήματα ε, και σε σχέση με τα διαζύγια, διότι τα διαζύγια δεν είναι νόμιμα και υπάρχουν και μεικτοί γάμοι όπου προκύπτουν νομικά προβλήματα, προβλήματα διαζυγίου. Αναγκάζονται αρκετέ γυναίκε να πάνε σε μια χώρα του εξωτερικού για να πάρουν το διαζύγιο. Αυτά ήθελα να προσθέσω και σα ευχαριστώ. Ο Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Η κυρία Συγκλάρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Κορνίλσεν έδωσε μια λεπτομερή περιγραφή και βεβαίως αρκετές λεπτομέρειες δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση. Πήγα εκεί έτσι με πολύ ανοιχτό μυαλό. Δεν είχα επισκεφθεί το Ισραήλ καθόλου ούτε ως τουρίστρια και για πρώτη φορά επισκέφθηκα τη Γάζα και τη Ραμάλα. Ε, ίσως το ταξίδι ήταν πολύ φορτωμένο και θα ήθελα να δω περισσότερα στην πλευρά του Ισραήλ. Ε, το Ισραήλ βέβαια έκανε διάφορες προσβολές, τις οποίες, προσφορές συγγνώμη, τις οποίες απορρίψαμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δεν έλαβα ικανοποιητικές απαντήσεις από πολλούς ας πούμε για τα 300 εκατομμύρια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην Παλαιστινιακή Αρχή ιδιαίτερα στη Γάζα και σε ποιο βαθμό αυτά τα χρήματα δεν φτάνουν στα χέρια της Χαμάς είτε άμεσα είτε έμεσα. Ένα άλλο ενοχλητικό ήταν η συμμετοχή ενός μέλους η οποία έδειχνε να τα ξέρει όλα και να τα λέει όλα και φοβούμαι ότι εκεί είχαμε απλώς μια σπατάλη των χρημάτων των φορολογουμένων. Η, το ταξίδι στη Γάζα, πολύ ενδιαφέρον να δούμε την κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες στο να διευκολυνθεί και να εξασφαλιστεί καλύτερη εκπαίδευση. Ξέρουμε ότι πολλές τάξεις λειτουργούν σε containers. Θα ήταν καλό να έχουμε περισσότερο χρόνο στην επαφή μας με τις ε, ΜΚΟ. Ένα άλλο θέμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθούν είναι το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η παραβίαση και ξέρουμε ότι υπάρχουν σοβαρές παραβιάσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ουσιαστικά είχε ανάμειξη στο θέμα αυτό. Η, κάθε Άστον, ε, παραδείγματο χάρη, δεν απάντησε στην ερώτηση που έθεσε εγώ την περασμένη εβδομάδα για την ε, βία που ασκείται εις βάρος των γυναικών μέσα στις ίδιες τους οικογένειες από άνδρες και παιδιά. Δεν συζητήθηκε καθόλου. Και όταν θέσαμε το θέμα αυτό στις πέντε υπουργού, με κοίταξαν έτσι με περιέργεια και ε, όταν συζητάμε για, το, για θέματα αυτού του είδους σε επιτροπές όπως ε, η δική μας, πραγματικά πρέπει να είμαστε κατηγορηματικοί ε, στο να καταδικάζουμε τέτοια φαινόμενα ντροπή τα οποία συμβαίνουν στις κοινωνίες αυτές ο Πρόεδρος. Κανείς άλλος? Δύο λόγια κυρία, για την κυρία Σένκλερ. Υπάρχουν πράγματα τα, οποία δεν τολμούμε να μιλήσουμε. Δεν ξέρω αν ε, είχατε την ευκαιρία να δείτε μια ταινία που βγήκε πρόσφατα στις οθόνες των κινηματογράφων. Ε, το γουρούν της Γάζας συγκεκριμένα λέγεται. Ε, είναι έτσι μια διασκεδαστική ταινία, μια κομμωδία θα έλεγα, αλλά Έχω πάει πολλές φορές στη Γάζα, στη λωρίδα της Γάζας και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι όλα όσα λέγονται σε αυτή την ταινία, έστω και με τρόπο έτσι αστείο, είναι αληθινά. Πήγα να το δω έτσι από περιέργεια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είδα κανένα λαθασμένο στοιχείο, κανένα λάθος στην παρουσία της πραγματικότητας. Και να πω ότι σε αυτή την ταινία υπάρχει μια σκηνή ε, σχετικά με το Βιάγκρα Και μπορώ να σας βεβαιώσω ότι έχω μιλήσει με γυναίκες στη Γάζα. Το Βιάγκρα είναι ένα προϊόν το οποίο περνάει από τα τούνελ, διακινείται πάρα πολύ στη λωρίδα της Γάζας. Και γιατί οι άντρες είναι πολύ συχνά σε άνεργοι, ε, βαριώνται και κάνουν ό,τι μπορούν. Ε, και αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν πάρα πολύ το Viagra. Ε, είναι μια πραγματικότητα την οποία ζουν οι γυναίκες καθημερινά μέσα σε αυτό το γκέτο στο οποίο έχει καταλήξει να είναι η λωρίδα της Γάζας. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Ας τελειώσουμε και αυτό το σημείο για να περάσουμε στο σημείο 9. Ε, αποστολή επίσκεψη στην Κοπενχάγη. Αντιπροσωπή τη Επιτροπή Δικαιωμάτων Γυναικών στην Κοπενχάγη. Ε, δύο ήμασταν. Ε, εγώ ήμουν ε, ένα, από τα δύο μέλη και δύο άντρε ήμασταν. ο κύριος Ταραμπέλα και εγώ ίδιος. και ε, συναντηθήκαμε μάλιστα και με τον Υπουργό τη Δύο Φίλων των που είναι επίσης άντρας. Ο κύριο Σορίν συγκεκριμένα. Ήταν πολύ αστείο. Ήμασταν τρει άντρε, μιλούσαμε για την ισότητα δύο φίλων. Συναντήσαμε βέβαια και τον Υπουργό Απασχόληση τη Δανία την ίδια ακριβώ μέρα. την Υπουργό μάλλον, την κυρία Φρέντριξεν. Ε, συναντήκαμε και με την μόνιμη Επιτροπή Ισότητας των Ιωφύλων που είναι πολύ καινούρια. Πρόσφατα δημιουργήθηκε. Ε, ακόμα και τα μέλη της είναι καινούργιοι βουλευτές. Συναντηθήκαμε με εκπροσώπους του Δήμου της Κοπενχάγης επίσης και με οργανώσεις της ε, κοινωνίας των πολιτών γυναικείες ε, φεμινιστικές οργανώσεις κλπ. Ε, η επίσκεψη αυτή διεξήχθη για να διαπιστώσουμε πού βρίσκονται τα δικαιώματα της γυναίκας και η κατάσταση των δύο φίλων στη Δανία. και επίσης να δούμε και τις προθέσεις της ε, προεδρία τη Δανίας για το επόμενο εξάμεινο. από ό,τι φαίνεται η Δανέζικη Προεδρία ενδιαφέρεται Δεν υπάρχει κάτι πολύ σαφές ακόμα στο πρόγραμμα της ε, Δανέζικης Προεδρίας αλλά κοιτάνε με πολύ θετικό μάτι το όλο ζήτημα. Αυτά συνοπτικά σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή σας για αυτή την επίσκεψή μας. Ε, μόνο εγώ εκ των παρόντων ήμουν εκεί, δεν ξέρω αν έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο. Εν πάση περιπτώσει θα τα δείτε όλα γραμμένα στην έκθεσή μας. Διαβάστε την. Ωραία. Κλείνουμε και αυτό το ζήτημα. Περνάμε στο 10. Μελέτη σχετικά με τις πτυχέ που σχετίζονται με τη ισότητα ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεση. Το 2010 η Επιτροπή υιοθέτησε μια έκθεση για, την, ε, για τις πτυχές ισότητας ε, της οικονομικής κρίσης. Η... Αποφασίσαμε ότι χρειαζόμαστε μια σε βάθος ε, ανάλυση αυτού του ζητήματος ε, απευθυνθήκαμε στο Ίδρυμα Μπροντολίνη. Η κυρία Λιμπεράκη είναι μαζί μας για να μας παρουσιάσει αυτήν την έκθεση. Έχει το λόγο. Okay. Thank you very much. I'm gonna be... Θα είμαι πολύ σύντομη. Δεν θέλω να σας κουράσω. Ε, θα διατρέξω τις διαφάνειες και θα αφήσουμε λίγο χρόνο και για συζήτηση, ελπίζω. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας υπενθυμίσω είναι ότι αυτή η έκθεση υποβλήθηκε τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους. Αυτό σημαίνει ότι σε εκείνη τη φάση είχαμε, είχε ξεκινήσει, μάλλον φαινόταν να έχει τελειώσει η αρχική η πιστοτική ασφυξία το πρώτο επεισόδιο ε, και ότι περνούσαμε σε μια φάση ανάκαμψης. Όμως υπήρχαν ενδείξεις για αυτό που ακολούθησε που πιο συγκεκριμένα ήταν το δεύτερο ε, και πιο ισχυρό επεισόδιο της κρίσης που είναι η κρίση του κρατικού χρέους. Συνεπώς η έκθεση καταγράφει τις εξελίξεις στο μέσον της εξελισσόμενης κρίσης. Το πρώτο τμήμα θα αναφερθώ στην κρίση σε σχέση με την ισότητα των δύο φύλων. Στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασής μου ε, προβλέψεις για το πρώτο τρίμηνο του 2011 πολιτικές, στατιστική ανάλυση και τέσσερις ε, ε, συγκεκριμένες μελέτες και στο τρίτο τμήμα της παρουσίασής μου για, τις, για τους κινδύνους και τα, τις πολιτικές και τα μαθήματα για το μέλλον. Λοιπόν, τι ξέρουμε για αυτή την κρίση. Η κρίση αυτή είναι καταρχήν διαφορετική από προηγούμενες κρίσεις είναι διαφορετική ως προς το, στη διάρκεια της, ως προς ε, την ισχύ της ε, και ως προς τις επιπτώσεις της ιδιαίτερα στα δύο φύλλα. Ξεκίνησε το 2008 ως πιστοτική ασφυξία εξαιτία ε, του, του, τομέα, του χρηματοπιστωτικού τομέα, αλλά το 2010 πλέον είχε μεταμορφωθεί σε μια κρίση σχετική με τα δημόσια οικονομικά και το κρατικό χρέος. Τρία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που την ξεχωρίζουν από προηγούμενες. Πρώτον, οι γυναίκε είναι πλέον πιο ενσωματωμένε στην αγορά εργασία, συνεπώ έχουν πιο πολλά να χάσουν σε σχέση με παλιότερε κρίσει. Δεύτερον, οι γυναίκε ήδη ζουν στο πετσί του αρνητικέ επιπτώσει με αύξηση τη ανεργία, αλλά αυτό που διαφάνηκε πλέον είναι ότι περνώντα στη δεύτερη φάση τη κρίση, δημοσιοοικονομικών και κρατικού ε, βλέπουμε ότι οι γυναίκες μπορεί να πληγούν ακόμα περισσότερο. Τρίτο χαρακτηριστικό που διακρίνει αυτή την κρίση από προηγούμενες ε, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές ε, ε, το mainstreaming και γενικότερα η διάσταση τη, του φύλου έχει πιο πολύ ενταχθεί στις ε, πολιτικές και γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες έχουν να χάσουν πιο πολλά, έχουν πιο πολλά να χάσουν από αλλαγές σε πολιτικές όπως ε, μείωση κοινωνικών δαπανών, ε, μείωση επενδύσεων σε ε, υποδομές κλπ. Η βασική ιδέα ε, και μήνυμα αυτή τη έκθεση είναι ότι οι γυναίκε είναι μια ένας ανεκμετάλλευτος πόρος ε, που θα μπορούσε να μας βοηθήσει να βγούμε από την κρίση και να εξασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη ευημερία. Η οικονομική ανάλυση βασισμένη σε, παλιότερες, σε προηγούμενες παρατηρήσεις προβλέπει ε, διάφορα σενάρια για το μέλλον. Πρώτο, Τη αργυρή εσωτερική επένδυση φόδρα να το πούμε, ε, με την έννοια ότι ε, πολλές δουλειέ γυναικών είναι προστατευμένες διότι αφορούν πιο μονομένα επαγγέλματα που δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από την κρίση. Με αυτή την έννοια ε, κινδυνεύουν λιγότερο. Δεύτερον, το σενάριο τελευταίος μέσα πρώτος έξω, «Λίφο», last in first out είναι αυτές που προσελήφθηκαν τελευταίες, συνεπώς ενδεχομένως είναι αυτές που πρώτες θα απολυθούν. Τρίτο σενάριο είναι το σενάριο FIFO, first in, first out. Αυτός που πρώτος ήρθε ε, ε φεύγει πρώτος. Ε, επειδή ε, οι γυναίκες αμείβονται λιγότερο, γίνονται πιο ελκυστικές και στην απόλυσή τους. Οπότε ε, ενδεχομένως μπορεί να συμβεί και αυτό. Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην, ε, στον, ε, στην εργασία υπάρχουν δύο δυνατότητες, δύο σενάρια. το σενάριο του αποθαρρυμένου εργαζόμενου που σημαίνει ότι επειδή δεν υπάρχουν πολλές θέσεις εργασίας οι γυναίκες βγαίνουν από την αγορά εργασίας ή το αντίστροφο, το αποτέλεσμα του πρόσθετου εργαζόμενου, επειδή ακριβώς τα νοικοκυριά αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, πολλές γυναίκες ενδεχομένως θα μπουν στην αγορά εργασίας για να βρουν απασχόληση. Και σε αυτή την ε, υφεσία, όπως και σε προηγούμενες, πολύ συχνά βλέπουμε και, τις, και τα δύο αυτά σενάρια και τις δύο αυτές τάσεις, ανάλογα με τη χώρα και ανάλογα με την πληθυσμιακή ομάδα. Παλιότερες μελέτες υποδεικνύουν ότι σε προηγούμενες περιπτώσεις ύφεση ε, οι γυναίκες είχαν επηρεαστεί λιγότερο από τους άντρες επειδή ακριβώς κάνουν διαφορετικά επαγγέλματα αλλά, αλλά η κρίση αυτή είναι πολύ πιο ισχυρή και, και βλέπουμε ε, ιστορικά ότι οι, οι φέσεις που είχαν παρελθεί πριν από 20 χρόνια ήταν λιγότερο ισχυρέ από τη σημερινή και από ό,τι αυτέ πριν από 5 χρόνια. Δηλαδή η ύφεση γίνεται όλο και πιο ισχυρή όσο περνάει ο χρόνο. Επίση, αυτή η ύφεση ε, είναι πιο επίμονη σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία ε, της ανεργίας. Και αυτό το έχουμε δει, θα τα δούμε τα στατιστικά στοιχεία. Ας δούμε το σημείο φετηρίας. Σημείο φετηρίας πριν την κρίση. Πριν την κρίση ε, είχαμε περισσότερες γυναίκες εργαζόμενες από ό,τι παλιότερα και από ό,τι τώρα, αλλά ε, με αμοιβή η οποία κειμενόταν. Οι γυναίκες ε, με, μικρό, με μικρά παιδιά είχαν χαμηλότερη αμοιβή από άλλες γυναίκες και μόνες γυναίκες ε, δούλευαν περισσότερο από τις άλλες μητέρες. Μόνες μητέρες ε, δούλευαν περισσότερο από άλλες μητέρες. Ε, οι γυναίκες γενικότερα ε, δούλευαν λιγότερο από τους ε, άντρες, δουλεύουν λιγότερο από τους άντρες, αμείβονται λιγότερο και ενδεχομένως εξαιτία των προηγούμενων δύο αλλά και για άλλους λόγους είναι πιο φτωχές από τους άντρες. Και αυτό κατά βάση παντού σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε, ας δούμε καταρχήν την εξέλιξη του ΑΕΠ από το 2007 μέχρι την αρχή του 2011. Ε, στην αρχή του 2011 φάνηκε να υπάρχει, να παρατηρείται μια ανάκαμψη, αλλά αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα. Η ε, η δεύτερη φάση της κρίσης ήταν πιο σαφή σε χώρες με προβλήματα στα δημοσιοοικονομικά τους όπως η Ιταλία ή η Ελλάδα αλλά αυτό το φαινόμενο άρχισε να γίνει πιο αφανής και στις άλλες ε, χώρες σιγά σιγά. Η ανάκαμψη δεν αύξησε την απασχόληση, αυτό είναι ενδιαφέρον φαινόμενο. Δηλαδή ήταν σαν να ήταν μια ανάπτυξη, μια ανάκαμψη χωρίς δημιουργία θέσεων εργασία. Και όπως σημαίνει στις περισσότερες υφέσεις, ε, οι διαφορές στην απασχόληση μεταξύ άνδρων και γυναικών δείχνουν να μειώνονται σε δείχνουν να μειώνονται σε όλη τη χώρα, σε όλες τις χώρες. Ε, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στην απασχόληση, οι γυναίκες φαίνεται όχι μόνο να διατηρούν τα ποσοστά τους, αλλά και να τα αυξάνουν. Οι άντρες φαίνεται ότι πλέονται περισσότερο από το φαινόμενο του ε, απογοητευμένου εργαζόμενου. Η συμμετοχή των γεγονών αυξάνεται κατά 1%, η συμμετοχή των ανδρών στην αγορά εργασία μειώνεται κατά 0,5%. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανεργία, παρόλο ότι η απώλεια θέσεων εργασία συγκεντρώνεται στις παραδοσιακούς ανδρικούς τομείς δραστηριότητας, έχουμε δει συγκρίσιμα νούμερα απώλειας θέσεων εργασία και για τις γυναίκες. Όμως, επειδή η ανεργία των ανδρών ήταν στην αρχή της κρίσης πολύ χαμηλότερη, η αύξηση, η ποσοστία αύξηση ε, ήταν θεαματική. Γι' αυτό το λόγο είναι πιο ε, προφανής από πλευράς δημοσιογραφικής κάλυψης. Αλλά βέβαια και για αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι τα στατιστικά στοιχεία για την απώλεια θέσεων εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι παρόμοια. Απλά οι, γυναίκες, οι άνδρες ξεκίνησαν από πολύ χαμηλά ποσοστά ανεργίας και γι' αυτό λόγο για αυτούς είναι πιο θεαματική η αύξηση της ανεργίας. Οπότε ε, δεν σας παρουσιάζω τις λεπτομέρειες. Να σας πω απλώς ότι στην αρχή της κρίσης οι τομείς, ε, οι πιο ανδρικοί τομείς επλήγησαν περισσότερο και αυτό στις περισσότερες χώρες. Η δεύτερη φάση της κρίσης όμως θα πλήξει πολύ, πιο πολύ τις γυναίκες μάλλον γιατί οι γυναίκες ε, αναλογικά αντιπροσωπεύονται περισσότερο στον κρατικό τομέα και τις κοινωνικές υπηρεσίες που θα πληγούν περισσότερο στη δεύτερη φάση και γιατί οι γυναίκες είναι επίσης οι κύριοι χρήστες των κοινωνικών υπηρεσιών και δικαιούχοι πολλών κοινωνικών παροχών. Τρεις λόγοι λοιπόν ε, θα ε, υπάρχουν που μας πείθουν ότι η δεύτερη φάση θα πλήξει περισσότερο τις γυναίκες. Παρόλο ότι τα στοιχεία που είχαμε μέχρι την αρχή του 2011 δεν καταγράφουν τέτοια αύξηση στην ανεργία των γυναικών. Ε, αυτοί οι παράγοντες οποίους σας ανέφερα αναπτύχθηκαν και θα εξακολουθούν να αναπτύσσονται αργότερα. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να περιμένουμε αύξηση των προβλημάτων ανεργίας στις γυναίκες. Τώρα, οι νέες φαίνεται να είναι πιο ευπαθείς από τις μεγαλύτερες και γενικότερα οι νέοι από τους πιο ηλικιωμένους. Οι άνω των 50 δείχνουν να εργάζονται για πιο πολύ χρόνο και δεν δείχνουν να πλήττονται περισσότερο από την ανεργία. Δηλαδή, μάλιστα, η συμμετοχή στην αγορά εργασία φαίνεται ότι αυξάνεται. Η αγορά εργασίας όμως ε, δεν είναι ομοιογενής. Ε, διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες έχουν διαφορετική πρόσβαση σε προνόμια για προστασία και παρόλο που η πλειοψηφία των εργαζόμενων στον, το δημόσιο τομέα είναι γυναίκες. Οι γυναίκες είναι ε, πλειοψηφία και στις ομάδες που εργάζονται χωρίς ε, κοινωνική προστασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τάσεις για τις πολιτικές. Ε, το, το περιβάλλον ασκεί πολλές αόρατες πιέσεις στην, στην ισότητα μεταξύ των και γυναικών. Πρώτον, εξαιτίας δημοσιονομικών λόγων, πρακτικά δεν υπάρχει ε, ειδικό σχεδιασμός για τις γυναίκες. Ε, θα μπορούσαμε να επηρεάσουμε τις γυναίκες μόνο όταν αφού αποφασίσουμε τις περικοπές ε, δούμε πώς θα τις εφαρμόσουμε και αν θα τις εφαρμόσουμε περισσότερες γυναίκες ή λιγότερο. Ε, επίσης, η παραγωγικότητα ε, δεν αφορά μόνο τα άτομα αλλά και τους τομείς. Στο μέτρο που οι γυναίκες εστιάζονται πιο πολύ σε δουλειές χαμηλής παραγωγικότητας, με χαμηλή αμοιβή, οποιαδήποτε σύνδεση ανάμεσα στην ατομική επίδοση και παραγωγικότητα και το, την αυξημένη ε, αμοιβή ή προστασία ε, είναι εκτός πραγματικότητας. Um, τώρα, φαντάζομαι ότι το βασικότερο πρόβλημα όσον αφορά τις πολιτικές, αν δούμε τις στατιστικές αναλύσεις και τα σχετικά ευρήματα, όπως εντοπίστηκαν στην έκθεση, είναι ότι υπάρχει ψυχασμός. Δηλαδή να πούμε, εντάξει, ναι, η κρίση είναι ένα πολύ ατυχές γεγονός, όλοι πλήττονται από την κρίση, αλλά υπάρχει αίσθηση ότι δεν είναι οι γυναίκες που είναι το επίκεντρο, αν θέλετε, στο μάτι του κυκλώνα. Αυτό θα έλεγα ότι δεν είναι ορθό, γιατί ο λόγος πρώτα απ' όλα είναι αναλυθές. Ε, η ανεργία των γυναικών δεν είναι τόσο ορατή όπως η ανδρική ενεργεία, γιατί εργάζονται σε άτυπες μορφές εργασίας, γιατί εργάζονται σε μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, είτε γιατί εργάζονται ε, σε μερικές επασχόλες κτλ και γιατί δεν είναι τόσο καλά ενταγμένα στα αγορά και πολύ απλά δεν καταγράφονται ως άνεργοι και άρα δεν καταγράφονται και ως υψηλό επίπεδο στις κοινωνικές παροχές. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο είναι εσφαλμένη αυτή η προσέγγιση είναι ότι ο υφεσυχασμός δίνει λανθασμένο μήνυμα όσον αφορά τις ε, πολιτικές. Δηλαδή αν δεχτούμε το γεγονός ότι για να βγούμε από αυτή την κρίση και να δημιουργήσουμε ευημερία για τις μελλοντικέ μας κοινωνίες, για άνδρες και γυναίκες εδώ στην Ευρώπη, θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε πλήρως τον εκμετάλλευτους πόρους που μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες στην εργασία. Δηλαδή, αν αφήσουμε πραγματικά στην άκρη και αν, ε, αγνοήσουμε, αν θέλετε, τη διάσταση του φύλου και βάζουμε σε γενικού στόχου από το 75% του πληθυσμού να απασχολείται ενεργά και να είναι οικονομικά ενεργή, χωρίς όμως να στοχεύουμε στο φύλλο και να μην υπάρχει ισότητα, τότε μπορούμε να καταλήξουμε σε άντρες με πολλές θέσεις εργασίας και γυναίκες με καμία θέση εργασίας. Και άρα ε, συνολικά μπορεί να επιτύχετε το στόχο ή να επιτύχετε και δεύτερο εισόδημα για κάθε νοικοκυριό. Το θέμα είναι η, η κατανομή ανάμεσα άνδρες και γυναίκες και θα δούμε ότι ο επιμερισμός θα είναι πολύ α, άνισος. Ένας άλλος κίνδυνος που δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε είναι ότι να επανέλθουν και πάλι στο προσκήνιο και πολύ έντονο τόσα στερεότυπα. Ε, το γεγονό ότι οι πραγματικοί εργαζόμενοι είναι άνδρε τελικά. Και όταν είναι λίγε τι εργασίε, οι άντρε θα πρέπει να ε, έχουν τη δουλειά και οι γυναίκε να πάνε παραδοσιακά και να κλειστούν στο σπίτι τους. Μπορεί να ακούγεται γελία ως απόψε και μόνο που το λέω, αλλά στην πραγματική ζωή και στις διάφορες έρευνες αξιών που ε, υπάρχουν και έχουν γίνει, βλέπουμε ότι είναι ιδέες που τελικά κερδίζουν έδαφος παντού στην Ευρώπη και παντού θα έλεγα στον ανεπτυγμένο κόσμο. Άρα, είναι πρόβλημα να μην δίνουμε έμφαση σε αυτή την ανάγκη να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε περαιτέρω την επίτευξη των στόχων της ισότητας ανδρών και γυναικών και σε παιδαπασχόλησης και οικονομικής ανεξαρτησίας. Ιδάλω θα καταλήξουμε σε καταστάσεις που θα μας θυμίζουν πολύ παλαιές εποχές. Και είμαι σίγουρη ότι αν τελικά πάμε τόσο πίσω, ότι ο δρόμος προς την ευημερία και το ενδεχόμενο εξόδου αυτή τη φοβερή κρίση θα ε, μειωθεί σημαντικά. Τα γενικά τώρα συμπεράσματα, ποια θα πρέπει να είναι. Η κρίση εμφανίστηκε σε δύο φάσεις. Με μία αδύναμη ανάκαμψη στο μεσοδιάστημα. Η πρώτη φάση ήταν μια ξεκάθαρη ε, κρίση ε, που θυμίζει σε μεγάλο βαθμό προηγούμενες επιπτώσεις που είχαμε σε θέματα ισότητας φύλων, αλλά το δεύτερο μέρος, η δεύτερη της κρίσης, που είναι μια πλέον καθαρά ε, κρίση δημόσιου χρέους, δίνει μια απόλυτη βεβαιότητα ότι οι περικοπές δημόσιες δαπάνες θα ζημιώσουν πολύ περισσότερο τις γυναίκες, ε, τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και τα ευάλωτα νοικοκυριά είναι αυτοί που κατά κύριο λόγο θα αισθανθούν περισσότερο αυτές τι αρνητικές συνέπειες. Οπότε παρότι τα στατιστικά ευρήματα έως τις αρχές του 2011 δηλώνουν ότι η πρώτη φάση είχε παρόμοια αποτελέσματα όπως προηγούμενες ε, περιπτώσεις ύφεσης, σε γενικές γραμμές όμως καταδεικνύει ότι στο δεύτερο σκέλος αυτής της κρίσης τα πράγματα δείχνουν πολύ πιο ζωφερά για το σύνολο της κοινωνίας βεβαίως, αλλά και ειδικότερα για τις γυναίκες. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι η ισότητα των φίλων δεν είναι ένας μεταξύ πολλών στόχων. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο σκεφτόμαστε όταν έχουμε την πολυτέλεια να δαπανίσουμε χρήματα. Και εκεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι κοινωνίες που θα απευθυνθούν περισσότερο με την κατανομή, πιο ε, ισότιμη κατανομή χρημάτων και εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, είναι αυτές που έχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν βήματα πίσω, έχουν δηλαδή μεγαλύτερο πρόβλημα στην ανταγωνιστικότητά τους και άρα είναι οι πρώτοι, αν θέλετε, ύποπτοι να εγκαταλείψουν το θέμα της των φίλων στην άκρη. Θέλω να επισημάνω τέσσερις κινδύνους που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρώτος είναι εξή. Επειδή η ανεργία των γυναικών και οι συνθήκε που του χαρακτηρίζουν στην αγορά εργασία είναι λιγότερο ορατοί παράγοντε, υπάρχει ο κίνδυνο να υποβαθμιστεί ε, ο ευάλωτο ρόλο των γυναικών και οι αρνητικέ συνέπειε αυτέ. Επίση, να δημιουργεί σύγχυση στι προτεραιότητε, πολιτικέ προτεραιότητε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το βασικό είναι ο άντρα που φέρνει, αν τα λεφτά στο σπίτι να έχει εργασία. Επίσης, ένας άλλος κίνδυνος είναι να θεωρούμε ότι η ισότητα των φύλων είναι μια πολιτική μόνο για τους καλούς καιρούς, οπότε τα αφήσουμε τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα. Αυτό θα ήταν καταστροφικό, πιστεύω, για τις προοπτικές της Ευρώπης και την έξοδο της από την κρίση. Τρίτος κίνδυνος. Οι χώρες που ανέφερα και πριν, που έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να κάνουν βήματα πίσω στην πολιτική ισότητα των φύλων, είναι οι χώρες εκείνες όπου η, η ισότητα μεταξύ των φύλων είχε δώσει τα πιο μακροχρόνια, αν θέλετε, ωφέλη. Εκεί λοιπόν όπου η συμμετοχή των γυναικών είναι λιγότερο ολοκληρωμένη, όσον αφορά τους όρους ε, αμοιβή και απασχόλησης, είναι πιο πίσω. Και ο τέταρτος κίνδυνος είναι η απουσία πληροφόρησης, ενημέρωση για θέματα φύλου, ειδικά όπου υπάρχει αποκεντρωμένη δικασία λήψη αποφάσεων, όπου η αρχή της επικουρικότητας ε, ισχύει και αυτό μπορεί να λειτουργήσει σωρευτικά. Δηλαδή όταν αυτά τα στοιχεία ε, εμφανιστούν μπροστά μας θα είναι πολύ αργά για να αντιμετωπίσουμε το γεγονός. Και δεν πρέπει να περιμένουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Οπότε κλείνοντας λέμε ότι η κρίση μπορεί να αποτελέσει καταλήτη για την πρόοδο, αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει και μια εύσχημη δικαιολογία για να αρνηθούμε την πρόοδο. Το τι θα γίνει τελικά εξαρτάται από τους πολιτικούς ηγέτες. Γι' αυτό και δεν θα πρέπει να υπάρχει εφησυχασμός. Και βεβαίως η μακροπρόθεσμη πρόοδο δεν θα πρέπει να θυσιαστεί στον βωμό των βραχυπρόθεσμων σκοπιμοτήτων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εισήγησή σας και την εισαγωγή που έγινε στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας που είμαστε ευτυχείς που συντάξατε την έκθεση αυτή, δεδομένου ότι χρειαζόμαστε κάποια στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ε, ισότητα και είναι χρήσιμο να βλέπει κανείς πώς η κρίση επηρεάζει τις γυναίκες. Αν κανείς δεν έχει μια συγκεκριμένη στρατηγική ε, σχετικά με την ισότητα των δύο φύλων και αντίστοιχα στατιστικά στοιχεία, δεν είναι δυνατόν να αναπτύξει πολιτικές. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ χρήσιμη η ερώτηση. Έχω δύο ερωτήσεις ή μάλλον ένα σχόλιο και μία ερώτηση. Μιλούμε για την όλη ιστορία της λιγότερης εργασίας. Κάζω ότι αναφέρεστε σε πληρωμένη εργασία ότι οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο ε, για πληρωμένη εργασία διότι αν κανείς συγκρίνει τη δουλειά των γυναικών και των ανδρών σίγουρα οι γυναίκες δουλεύουν πολύ περισσότερο αλλά η πληρωμένη εργασία ε, των γυναικών είναι λιγότερη. Και όταν μιλούμε για τις προοπτικές ανάπτυξης Ε, υπάρχουν διάφορες δυνατότητες. Από τη μια είναι η πτυχή κοινωνική. Η γυναίκα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Από την άλλη, αν θέλουμε ανάπτυξη, η γυναίκα πρέπει να είναι παρούσα στην αγορά εργασίας για να παραγάγει, για να αποδώσει. Εικάζω λοιπόν ότι αναφέρεστε σε πληρωμένη εργασία, όταν λέτε ότι οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο. Άρα λοιπόν υπάρχουν κοινωνικοί λόγοι αλλά και οικονομικοί λόγοι ώστε να αυξηθεί ο ρόλος της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Ενώ από την άλλη υπάρχει το θέμα της παραγωγικότητας. Όπως είπατε, οι γυναίκες συχνά δουλεύουν σε κλάδους, σε τομείς όπου είναι δύσκολο να αυξηθεί η παραγωγικότητα. Πρόκειται για απασχόληση στην οποία κυριαρχούν οι γυναίκες. Όταν κανείς συγκρίνει παραδείγματος χάρη ένα νηπιαγωγείο με, και την παραγωγικότητα σε αυτό με μία μονάδα κατασκευής αυτοκινήτων. Ε, δεν, μπορεί, δεν είναι δυνατόν να γίνει σύγκριση. Όταν λοιπόν κανείς δουλεύει ε, σε ένα νηπιαγωγείο για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η παραγωγικότητα τι πρέπει να κάνει κανείς, δηλαδή να αλλάζει δύο φορές παραπάνω τα, τα πάμπερς των παιδιών ή να μαθαίνει διπλάσια γνώσεις τα παιδιά. Αν θέλει, ας πούμε όταν παίζει κανείς ένα συμφωνικό έργο θα το παίξει δύο φορές πιο γοργά, πιο γρήγορα το κομμάτι αυτό και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει την παραγωγικότητα δεν είναι δεν είναι λογικό αυτό. Παρακαλώ, έχετε το λόγο τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ, όπως και εσείς υπογραμμίσατε, εκτιμώ ιδιαίτερος τη μελέτη αυτή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και σημαντική, δεδομένου ότι έχουμε αυτή τη στιγμή στατιστικά στοιχεία σε την περίοδο κρίσης. Αρχίζω από το πρώτο σημείο που υπογραμμίσατε και που και μένα μου προκάλεσε μεγάλη απορία η ιδέα η οποία επικρατεί και εξελίσσεται ότι σε περίοδους κρίσης θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στους άνδρες να βρουν εργασία. Στη χώρα μου υπάρχει μια μελέτη του Μαρτίου και πάνω από το 60% των ανδρών θεωρούσαν ότι σε περίοδους κρίσης οι άνδρες έπρεπε να έχουν προτεραιότητα στην απασχόληση. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα στερεότυπα επανεμφανίζονται, επαναγεννώνται σε περιόδους κρίσης. Συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέτε. Είναι πολύ σοκαριστικό αυτό. Και εναντίον αυτής της νοοτροπίας πρέπει να αγωνιστούμε. Βέβαια, πρόκειται για στερεότυπα που είναι πολύ δύσκολο να τα καταπολεμήσει κανείς, διότι είναι καλά ριζωμένα στον πληθυσμό. Δεύτερο σημείο επί του οποίου θα ήθελα να αναφερθώ. Όλοι σε επίπεδο Ευρώπης, κρατών, οικογένειας έχουμε επενδύσει πολλά και πολύ στην ίση εκπαίδευση και κατάρτιση αγοριών και κοριτσιών και τα κορίτσια στην εκπαίδευση, στις εξετάσεις ε, αποδίδουν εξίσου καλά ή και καλύτερα. Και γι' αυτό θεωρώ πολύ σοκαριστικό το δεύτερο σημείο, ότι στη συνέχεια δεν βρίσκουν την ίδια ισότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Και δεν υπάρχει η ίδια ελπίδα καριέρας, ούτε και τα ίδια επίπεδα μισθών. Και όπως έλεγε και ο αξιότιμος πρόεδρος προλίγου σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσχέρειας οι χώρες, τα κράτη θέλουν ας πούμε να οθήσουν όλες τις δυνάμεις στην αγορά εργασίας και βεβαίως οι γυναίκες αποτελούν στον ίδιο βαθμό κομμάτι αυτού του δυναμικού. Άρα λοιπόν πρεσβεύουμε και υποστηρίζουμε την ε, ισότητα στη μόρφωση αγοριών και κοριτσιών αλλά όλα όσα περιορίζουν την πρόσβαση της γυναίκας στην αγορά εργασίας λειτουργούν ως ανασταλτικός παράγων ε, και, ε, και μάλιστα μεγαλύτερος, λειτουργούν ως μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγων σε περίοδους κρίσης. Πολύ σωστά η μελέτη σας καταδείχνει ότι η ανεργία των ανδρών είναι πολύ πιο ορατή από αυτή των γυναικών. Πριν από την κρίση ούτως ή άλλως δεν υπήρχε ισότητα και τώρα εν μέσω κρίσης η απόσταση αυτή μεταξύ των δύο μεγαλώνει. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν μέτρα για να βγούμε από την κρίση και για να αναπτυχθεί η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Γουμάη. Ευχαριστώ, αγαπητέ Πρόεδρε. Σε ευχαριστούμε, Αντιγόνη, για τη θαυμάσια δουλειά και δεν έχω αμφιβολία ότι Ε, ε, ε, είπα στη συζήτησή μας ότι η κρίση αυτή έπληξε τους, τους άνδρες, τον κατασκευαστικό τομέα, τον οικονομικό τομέα. Αν οι Lehman Brothers ήταν, δεν ήταν brothers αλλά sisters, ίσως δεν θα προέκυπτε η κρίση αυτή. Στον πρώτο κύκλο λοιπόν της κρίσης επηρεάστηκε η απασχόληση των ανδρών ακριβώς επειδή σε αυτούς τους τομείς κυριαρχούν οι άνδρες. Από την άλλη, δεν λάβαμε σοβαρά υπόψη το δεύτερο κύκλο. Στο δεύτερο κύκλο που επηρεάζει πολύ περισσότερο τις γυναίκες, διότι αυτές έχουν ε, βραχυπρόθεσμα συμβόλαια, ε, ή δεν έχουν πλήρη απασχόληση κλπ. Πράγματι λοιπόν χρειαζόμαστε στατιστικά στοιχεία για αμφότερα τα φύλλα και υπάρχει μια δυναμία στη στρατηγική του 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν, υπάρχει μόνο ένα στοιχείο, ότι συνολικά θέλουμε 75% απασχόληση στο πλαίσιο αυτό. Ενώ η στρατηγική της ε, Λισαβόνας έλεγε ότι οι γυναίκες πρέπει να περάσουν από το 50% στο 60%, οι άνδρες από το 60% στο 70% κλπ. Εγώ βεβαίως πιστεύω στην ισότητα των δύο φύλων και κατανοώ ότι όσο μεγαλύτερη ισότητα φύλων έχουμε, τόσο μικρότερη κρίση. Αν όσο καλύτερα κατανέμεται ο προϋπολογισμός, τόσο το καλύτερο για την ε, για την ισότητα και η απάντηση είναι περισσότερη δημοκρατία. Η απάντηση στην κρίση είναι ότι θέλουμε περισσότερη ισότητα. Πρέπει βέβαια να αλλάξει και η νοτροπία των ανδρών και χαίρομαι που προλίγου αναφέρθηκε ακριβώς αυτή η προκατάληψη ότι πρέπει σε περίοδο κρίσης να δοθεί προτερότητα στους άνδρες. Αλλά η αγορά εργασίας έχει αλλάξει πλέον. Δεν έχουμε μόνον τους ε, υπαλλήλους γραφείου και τους ε, χειρόνακτες και οι γυναίκες μπορούν να κάνουν αυτές τις δουλειές. Αυτή τη στιγμή έχουμε το 60% των γυναικών που εγκαταλείπουν το πανεπιστήμιο. Ως μητέρα δύο παιδιών, δύο αγοριών, ανησυχώ λίγο, αλλά ελπίζω ότι οι επόμενες γενιές θα τα καταφέρουν καλύτερα, με καλύτερη μόρφωση, με καλύτερους συντρόφους κλπ. Πιστεύω ακράδαντα ότι είναι κρίσιμη σημασίας η Κομισιόν όχι μόνο να ομιλεί περί ισότητας των δύο φύλων και περί ενσωμάτωσης της διάστασης της ισότητας παντού, αλλά και να δρά, να δρά. Και υπάρχει και ένας άλλος λόγος που τα λέω όλα αυτά. Κοιτάζοντας την κρίση βλέπει κανείς τις γυναίκες όλο και περισσότερο απελπισμένες και να, να τραβιούνται μακριά από την πολιτική και να εντάσσονται ή να υποστηρίζουν ε, εξτρεμιστικές απόψεις. Και αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Άρα λοιπόν όλοι μας στην αίθουσα αυτή θα πρέπει να μελετήσουμε αυτό το πολύτιμο έγγραφο αλλά να το πάρουμε και ως θετικό παράδειγμα ότι, και να πούμε ότι η κρίση δεν είναι μόνο δυσκολία αλλά και ευκαιρία. Είναι ευκαιρία να δώσουμε απάντηση στην κρίση, να συμπεριλάβουμε δηλαδή τις γυναίκες πολύ περισσότερο και στη λήψη αποφάσεων και στη δράση. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Στρέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω και εγώ με τις συναδέλφους. Συγχαίρω την κυρία Λιμπεράκη για αυτή την πολύ σημαντική μελέτη και πολύ επίκαιρη. Έχουν γίνει και άλλες μελέτες σε σχέση με το ρόλο, για παράδειγμα, των γυναικών, το ρόλο που οι γυναίκες δεν ανέλαβαν στην κρίση, γιατί οι γυναίκες δεν είναι υπεύθυνε για τη δημιουργία της κρίσης αυτής, είναι όμως τα βασικά θύματα της κρίσης. Και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, οι, οι Αμερικάνοι καλούν τις γυναίκες καλούσαν τις γυναίκες να διορθώσουν τα λάθη των ανδρών και την κρίση που είχαν δημιουργήσει στην αρχή της κρίσης αυτής. συνειδητοποιούμε ότι οι επιπτώσεις της κρίσης, ιδιαίτερα στη δεύτερη φάση της, θα είναι πιο... θα βαρύνουν πιο πολύ τις γυναίκες από τους άντρες. Στην πρώτη φάση η οικοδομή απασχόλησε πιο πολύ άντρες και ήταν αυτό ο τομέα που επλήγει καταρχήν και γι' αυτό το λόγο η γυναική ενέργεια δεν ήταν τόσο υψηλή. Στη δεύτερη φάση όμω. η κρίση συνδέεται πλέον με μια ε, οικονομική, με την οικονομική πτυχή ε, με περικοπές και αυτό θα επηρεάσει και τις γυναίκες. οι γυναίκες είναι οι τελευταίες που προσλαμβάνονται και οι πρώτες που απολύονται. Και αυτό γίνεται όλο πιο ορατό σε περίοδους κρίσης. Γιατί όπως είπε και η συνάδελφός μου, έχουμε και την αναβίωση ή την επιβίωση των στερεοτύπων στην κοινωνία μας. Παράδειγμα, πριν από λίγες μέρες έβαλα στο Twitter τη συζήτηση που κάνουμε και κάποιος απάντησε τι σχέση είχε κρίση με, τα, με, με τις γυναίκες και πώς είναι το να επηρεάζει διαφορετικά τις γυναίκες από τους άντρες. <laughs> δηλαδή κάποιοι θεώρησαν παράξενο να συζητούμε την κρίση υπό το πρίσμα του φίλου. Έχουμε λοιπόν πολύ μακρύ δρόμο μέχρι να αλλάξουν οι νοοτροπίες. Επίση να πω και το εξή. Τα project που χρηματοδοτούνται με μικροπιστώσει έδωσαν καλύτερα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, πάνω από το 90% από αυτά τα project έδωσαν θετικά αποτελέσματα ε, και τα περισσότερα από αυτά τα διαχειρίζονται γυναίκες. Και δεν επωφελούνται μόνο οι ίδιες, αλλά όλη η οικογένεια και κυρίως τα παιδιά τους. Σήμερα διάβασα μια είδηση που με εξέπληξε πραγματικά ότι εξαιτία της κρίσης των περικοπών, των... της οικονομικής δυσπραγίας, διάβαζα ότι παιδιά στην Ελλάδα λιποθυμούν στα σχολεία λιποθυμούν γιατί ε, δεν τρώνε αρκετά. Για παράδειγμα, τα τελευταία κρούσματα ήταν για παιδιά ε, που είχαν να φάνε δύο μέρες. Και όλα αυτά σε μια Ευρώπη ανεπτυγμένη, μια Ευρώπη της ευημερία. Ας σκεφτούμε λοιπόν τις συνέπειες της κρίσης πάνω στα παιδιά. Ε, τα επιπτώσεις στα παιδιά συνδέονται πολύ με τις επιπτώσεις της ίδια της γυναίκες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Λιμπεράκη, έχετε το λόγο για να συνοψίσετε. Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας και για την φιλική και θετική υποδοχή της μελέτης μας. Πιστεύω θερμά στην ανάγκη να έχουμε στοιχεία ε, αναλυόμενα αναφύλλω. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει σοβαρή συζήτηση. Είναι ντροπή να μην έχουμε ε, να ένα φύλλο στατιστικά στοιχεία μέχρι τώρα. Παρ' όλα αυτά, και κάνω ένα άλμα σε ένα διαφορετικό θέμα, τα στερεότυπα δείχνουν να είναι πολύ πιο παγιωμένα, πιο ριζωμένα από ό,τι κανείς θα ανέμενε. Είναι έτσι η φύση των πραγμάτων, τα στερεότυπα προφανώς αποθηκεύονται κάπου στο πίσω μέρος του μυαλού, πολύ βαθιά. Και χρειάζεται ε, για να, να, βγάλουμε το μέσα έξω, να τα φέρουμε όλα τα πάνω κάτω για να τα καταργήσουμε τα στερεότυπα. Και γι' αυτό το λόγο ο κίνδυνος είναι μεγάλος. Υπάρχουν καλά νέα στο πεδίο της ισότητας των δύο φύλων. Σε όλο τον κόσμο. Ακόμα και στις πιο φτωχές χώρες. Βλέπουμε τουλάχιστον ενδιαφέρουσες εξέλιξεις. Όμως Πρέπει επίσης να πούμε ότι οι ιεραρχίες, οι προτεραιότητες, η συνείδηση ε, των κυβερνώντων επηρεάζονται πάρα πολύ από παλαιότερες αξίες και από ε, παλαιότερες κατανομές καθηκόντων μεταξύ άνδρων και γυναικών. Οπότε είναι πολύ πιθανό να δούμε ε, ε μισογενικές αξίες ε, που ως τώρα τις είχαμε βγάλει έξω από την πόρτα να μπαίνουν από το παράθυρο πλέον και από όλα τα παράθυρα ταυτόχρονα ενδεχομένως και ενδεχομένως και από την καπνοδόχο που κανένας δεν κοιτάει πολλές φορές. Προφανώς εννοούσα ότι οι γυναίκες δουλεύουν λιγότερο ως αμοιβόμενοι εργαζόμενοι. Προφανώς και γνωρίζω ότι δουλεύουν περισσότερες ώρες συνολικά από τους άντρες. Παρόλο ότι η περιπτωσιολογική μελέτη του Ηνωμένου Βασιλείου που συμπεριλάβαμε φαίνεται να δείχνει ότι η διαφορά στο συνολικό αριθμό ώρων εργασία, ε, και μη αμοιβόμενη, ανάμεσα στις γυναίκε και του άντρε, στην Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα δείχνει να μειώνεται. Πριν όμως αρχίσουμε να χειροκροτούμε τον Βασίλειο, να πω ότι ο λόγος είναι πως οι γυναίκες αφιερώνουν λιγότερες ώρες στον οικοκυριό τους και όχι γιατί οι άντρες αφιερώνουν περισσότερες. Ε, η διαφορά μπορεί να μειωθεί είτε με τις γυναίκες να μειώνουν την απασχόλησή τους με τον οικογενειό είτε με τους άντρες να την αυξάνουν. Ε, το πρώτο από τα δύο συμβαίνει. έχουμε κάποια καλά αποτελέσματα αλλά ας μην εφησυχάζουμε. Ακόμα και οι καλύτερες στατιστικές ε, αποκρύβουν κινδύνους. Χρειάζονται βαθιά μελέτη και ερμηνεία. Το θέμα της ορατότητας επίσης είναι πολύ σημαντικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Μιλώντας με καθημερινούς ανθρώπους και λέγοντάς τους ότι συζητούμε τις επιπτώσεις κρίσης την ισότητα των δύο φίλων ε, και μας λένε ότι τι ανοησία είναι αυτή και δεν καταλαβαίνουν γιατί θα πρέπει να υπάρχουν τέτοιες επιπτώσεις. Ε, το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι πολύ ορατό στον καθημερινό άνθρωπο. Ε, να τελειώσω κάνοντας το, την εξή παρατήρηση. Δεν εμπίπτουν όλες οι γυναίκες στην ίδια κατηγορία. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες γυναικών, διάφορες ομάδες γυναικών που επηρεάζονται από την κρίση με διαφορετικό τρόπο και σε διαφορετικές φάσεις. Από πλευρά προτεραιοτήτων θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τις πιο ευπαθείς ομάδες των γυναικών και μετά να περάσουμε στις υπόλοιπε. Και για να εξυπηρετήσουμε αυτές τις πιο ευπαθείς ομάδες γυναικών Μερικές φορές ε, πρέπει να είμαστε πολύ αποφασιστικοί και να αναθεωρήσουμε ενδεχομένως κάποια προνόμια ε, ομάδων είτε γυναικών είτε ανδρών είτε μεικτών ομάδων. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ χαρά μου που δούλεψα σε αυτή τη ε, μελέτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Ήταν μεγάλη χαρά και για μας ε, να σας έχουμε εδώ παρούσα και για την παρουσίαση της έκθεσής σας. Όπως ε, είπαν και οι συνάδελφοι και εγώ θεωρώ ότι είναι μια πολύ χρήσιμη έκθεση που συμβάλλει πάρα πολύ στην ε, τόσο επίκαιρη συζήτηση. Να αφήσουμε τώρα το σημείο 10 στην συνέντευξη, αλλά έτσι ολοκληρώνουμε και τις σημερινή μας εργασίες. Αύριο το πρωί στις 9 ξεκινούμε με τις ψηφοφορίες. στόχος είναι να ξεκινήσουμε 9 ακριβώς. Όχι 9 και 5, όχι 9 και 10, 9 ακριβώς. Λοιπόν, κλείνω τη συνεδρίαση για σήμερα και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9.